Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε. Λίγοι είμαστε προς το παρόν. Το ΕΛΚ όμως εκπροσωπείται σχεδόν, ε, ε, έχει μεταβεί σχεδόν αυτάνδρο στο Ελσίνκι. Αλλά και οι άλλοι έχουν κάποια σύνοδο κόμματος. Και έτσι δεν έχουμε τόσους σήμερα παρόντες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε και τη δουλειά μας σωστά. Και έτσι ξεκινώ με το σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης που είναι η έγκριση. Θέλετε να αλλάξετε κάτι, έχετε κάποια παρατήρηση, όχι. Εγκρίνεται λοιπόν, όπως έχει. Πρακτικά. Έχουμε το σχέδιο πρακτικών της 24ης Σεπτεμβρίου στο φάκελό σας. Παρατηρήσεις έχετε. Όχι. Όσοι ήθιστε λοιπόν προτείνω να θεωρηθεί πως έχουν εγκριθεί τα πρακτικά εφόσον δεν εγερθούν αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της τρέχουσας συνεδρίασης. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Η διερμηνία στις εξής γλώσσες γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, τσεχικά, εστονικά, ουγγρικά, πολωνικά, βουλγαρικά και ρουμανικά και ενημερώνω ότι όπως πάντα έχουμε web streaming μετάδοση από το διαδίκτυο της συνεδρίασης. Αυτά για τις ανακοινώσεις. Και περνώ αμέσως στο επόμενο θέμα της ημερήσης διάταξης, εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης για την απαλλαγή 2017, συνολικός προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κέντρο Μετάφρασης για τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον εισηγητή κύριο Στρογεύσκη, ο οποίος είναι παρόν, κατάθεση τροπολογιών έως τις 16 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, ψηφοφορία στις 21 Ιανουαρίου του 2019, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού στις 20 Φεβρουαρίου θα ψηφίσει τη δική της έκθεση. Έχουμε λοιπόν όπως και πέρσι αποφασίσει να μην περιοριστούμε μόνο στο γενικό σχέδιο του προϋπολογισμού αλλά να μιλήσουμε συγκεκριμένα και για το κέντρο μετάφρασης για τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη γνωμοδότησή μας. Γι' αυτό και παρακαλώ τώρα τον κύριο Στροιεύσκη να λάβει το λόγο για να μας παρουσιάσει τις ε, ιδέες του. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και καλημέρα σας. Αυτά τα δύο σημεία θα σας τα παρουσιάσω μαζί και πολύ συνοπτικά μάλιστα, γιατί από πολλές απο... Ε, απόψεις ε, ε, συνάδουμε με την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις. Σε ό,τι αφορά το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τις ε, ε, δικές μας παρατηρήσεις και αξιολογήσεις που επαναλαμβάνονται. Μερικές φορές είμαστε ικανοποιημένοι, μερικές φορές συγκρατημένα ικανοποιημένοι και μερικές φορές ε, δυσαρεστημένοι. Καταρχήν εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τα αποτελέσματα το προγράμματο Έρασμος. Πάνω από 1 εκατομμύρια φοιτητέ αποφελήθηκαν και σύντομα θα γίνουν 10 εκατομμύρια των φοιτητών ε, που θα δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια του Έρασμος και αυτό θα πρέπει να το γιορτάσουμε. Και μάλιστα δύο φορές ε, διευρύνθηκε το Έρασμος και μάλιστα ε, θα τριπλασιαστεί η ανάπτυξη του, κάτι που από την δική μας άποψη Επιτροπής Πολιτισμού είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτή η ενίσχυση του Έρασμος. Επίσης, ε, είχαμε εκτενή συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη και μάλιστα υπήρχε και διάσταση απόψεων, ε, γιατί ε, Ελήφθησαν ταυτόχρονα δύο αποφάσει της ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύη αφενός και αφετέρου της μείωσης του προγράμματος για τον εθελοντισμό των νέων. Η Επιτροπή Πολιτισμού, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στα θέματα αυτά, δεν επέτρεψε να δημιουργηθεί ένα κενό ε, για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οπότε και τα δύο προγράμματα προχώρησαν και ήδη δρέπουμε τους πρώτους καρπούς. Πάνω από 2.500 νέες θέσεις ε, έχουμε εργασίες για την τοποθέτηση νέων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Τρίτο στοιχείο που δυστυχώς ε, είναι προβληματικό ε, για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε χαμηλό βαθμό απορρόφησης ε, του προγράμματος ε, και Ευρώπη για τους πολίτες και για τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη Δημιουργική Ευρώπη και για την Ευρώπη για τους πολίτες έχουμε προβληματισμό γιατί την χαμηλά τα ποστά επιτυχίας των έργων και θα έπρεπε να ενταθεί ο ρυθμός και να έχουμε πολύ περισσότερα προγράμματα και επίσης επισημαίνουμε το ρόλο του εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευση οπτικοακουστικών μέσων και πολιτισμού στην υλοποίηση των τριών προγραμμάτων ε, για τα οποία είναι αρμόδιος και νομίζω ότι ε, η αξιολόγηση μας μπορεί να είναι θετική για το ρόλο του ΕΑΣΕΑ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Μεταφραστικό Κέντρο για τους ε, Οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρυσι το στοιχείο αυτό είχε εξεταστεί ξεχωριστά. Θα ήθελα να τονίσω ότι ε, ω συναρμόδιο για τον προπολογισμό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο επηρεάζει και την εκτέλεση του προπολογισμού. Γι' αυτό και κάνουμε κάποιε προτάσει. Ε, καταρχήν, ω Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, καλούμε την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, που είναι αρμόδια τη ουσία, να συμπεριλάβει τι προτάσει τη γνωμοδότησή μα. Καταρχήν, ε, εξακολουθούμε να είμαστε δυσαρεστημένοι από το επίπεδο εκτέλεσης των έργων και επίσης ε, θα διαπιστώνουμε ότι θα πρέπει να γίνουν σημαντικές διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσουμε σαφώς καλύτερη ποιότητα. Σε ό,τι αφορά την απαλλαγή για το ε, κέντρο, αυτό το κέντρο μεταφράσεων, θα πρέπει να Καταρχήν, να εκφράσουμε την ισχυρή δεσμευσή μα υπέρ τη πολυγλωσία. Αυτό μάλιστα φάνηκε και στη συζήτηση και τα σχόλια των Ευρωβουλευτών, γι' αυτό το τονίζουμε. Επίσης, έχουμε τη νέα τιμολογιακή δομή για τη μεταφρασία γράφων και μάλιστα χάρη σε αυτή τη νέα τιμολογιακή δομή, το 2017 είχαμε και αναβάθμιση της ποιότητας, αλλά και εξοικονομήσει, ενώ τα έσοδα δεν έχουν μειωθεί. Η εξοικονόμηση ανήρθε σε πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ μάλιστα. Επίσης, κατά τα τέλη του 2018 διαπιστώνουμε με ικανοποίηση ότι ε, ο αριθμός των πελατών του κέντρου ανήλθε στους 65, κάτι που δείχνει μια καλή δυναμική και πολύ θετική πορεία. Και τέλος, ενθαρρύνει το κέντρο να θέσει τη διάθεση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νέα έκδοση της διαδραστικής ε, βάσης ε, ονοματολογίας του ΙΑΤΕ που είναι πολύ σημαντικό να γίνει μέχρι το τέλος του 2018 εξασφαλίζονται στη συμπόρευση της διοργανικής βάσης δεδομένων ορολογίας με την καινοτομία. Και έχουμε έτσι κοινό παρανομαστή σε όλα αυτά τα θέματα. Χάρη στην ανανέωση του ΙΑΤΕ. Ευχαριστώ. Ja vielen Dank. Ευχαριστώ και εγώ. Πρέπει να περιμένω τελειώσει η διερμηνία τη φράση της. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την παρουσίαση της γνωμοδότησης. Οι σκιώδεις ηγητές, ο πρώτος ο Λουίτζι Μωράνο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Και θα είμαι λακωνικός. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο για την εξαιρετική βάση εργασίας που μας παρουσιάζει, αλλά και γιατί με πολύ εύστοχο τρόπο περιέγραψε τα κύρια ζητήματα που μας έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν αλλά και επανέρχονται με το αίτημα για επίλυση. Στα άλλα θέματα δεν θα επισέλθω, αλλά θα σταθώ στο ότι μειώνεται το συνολικό ποσοστό σφάλματος και το κρίνω αυτό ως θετικό μήνυμα γιατί φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε σοβαρά υπόψη και τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και βέβαια του Κοινοβουλίου, δηλαδή τις δικές μας για τα δικά μας θέματα. Επίσης καταγράφω κάποια ανησυχία σε σχέση με τους μηχανισμούς εταιρικού ελέγχου για το Erasmus Plus και το ε, Δημιουργική Ευρώπη που μέχρι τώρα δεν έχουν ε, ε, υλοποιηθεί, αλλά νομίζω ότι είναι ζητήματα αυτά που μπορούν εύκολα να επιληθούν. Ένα ζήτημα το οποίο μπορεί εύκολα να επιληθεί νομίζω είναι το έξω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πώ είναι πολύτιμη και για τη δική μα τη δουλειά η αιτήσει λογαριασμοί του ελεγκτικού συνεδρίου του, οι οποίοι όμω δημοσιεύονται πολύ συχνά με μεγάλη καθυστέρηση. Και έτσι δεν μπορούν να ληφθούν ε, υπόψη με τη δέουσα προσοχή παρά μόνο πολύ αργά. Και σε αυτό ε, θα ήθελα να σταθώ στο θέμα του Κέντρου Μετάφρασης για του Οργανισμούς και τι Υπηρεσίε Ευρωπαϊκής Ένωση, αλλά και στο θέμα των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Τρίπελ. Ευχαριστώ, Πέτρα. Δεν έχω πολλά να προσθέσω και εγώ ευχαριστώ το συντάκτη. Και όπως είπε και ο κύριος Μοργάνο, Για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι έχουμε πολύ επιτυχημένα προγράμματα, πολύ περισσότερο επιτυχημένα στο δικό μας από ό,τι σε άλλους τομείς, με πολύ καλύτερο ποσοστό υλοποίησης και μικρό ποσοστό σφάλματος, μειώνεται δηλαδή όπως είπες και εσύ Τζι και αυτό βέβαια το κρίνουμε θετικά, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ε, εκείνοι που διαχειρίζονται τα προγράμματα, είτε είναι οι υπηρεσίες, είτε είναι οι επιτόπου παράγοντες που τα διαχειρίζονται, κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και ε, γιατί αποδεικνύεται βέβαια ότι έχουν καλή υποδοχή τα προγράμματά μας, αλλά και γιατί εκτελούνται σωστά. Κάποια μικροπροβλήματα παραμένουν, αλλά όχι σοβαρά. Γιατί ξέρουμε ότι σε άλλους τομείς ε, το ποσοστό υλοποίηση, το ποσοστό εκτέλεση είναι πολύ διαφορετικό στα διευθυντικά ταμεία, παραδείγματι ορισμένων κρατών. Ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι χαοτική. Εμεί νομίζω ότι έχουμε καταφέρει αρκετά καλά, έω πολύ καλά. Και θα συμφωνήσω και με τον συντάκτη ότι σε μεγάλο βαθμό έχουμε να κάνουμε με υποχρηματοδότηση, έχουμε να αντιμετωπίσουμε υποχρηματοδότηση. Ακριβώς επειδή είναι τόσο καλή η εκτέλεση, το ποσοστό εκτέλεση, αν είχαμε περισσότερα χρήματα στη θέση μα, θα είχαμε και πολύ καλύτερα αποτελέσματα στου τομεί που μα ενδιαφέρουν τόσο πολύ. Εξού και πιστεύω ότι μπορούμε με την απαλλαγή αυτή και επί τη ευκαιρία τη αντιπαράθεση για το προσεχή πολίτε στο νομικό πλαίσιο να αποδείξουμε ότι η δική μα δουλειά είναι καλή δουλειά, είναι παραγωγική δουλειά και μπορούμε ε, να πούμε ότι έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα πέραν κάποιων μικροπροβλημάτων τα οποία όλες δεν μπορούν να αποδοθούν σε εμά. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω άλλον σκιώδη συγγητή εδώ, σκιώδη συντάκτη. Ε, Μια-δύο παρατηρήσεις θέλω και εγώ να κάνω. στο πρώτο υποσημείο της γνωμοδότησης όπου κάνετε λόγο για 9 εκατομμύρια φοιτητέ για τους οποίους εξασφαλίζεται η κινητικότητα. Θα ήθελα μια διαφορετική διατύπωση, σας παρακαλώ πολύ. γιατί έχουμε μπορέσει με το Εράσμους ε, ή έχουμε να αντιμετωπίσουμε και έχουμε αντιμετωπίσει με το Εράσμους και κάποιες ε, προκαταλήψεις ε, και έτσι έχουμε μπορέσει να ξεπεράσουμε την ιδέα ότι το Εράσμους είναι μόνο για τους φοιτητέ, αλλά έχουμε συμπεριλάβει και σπουδαστές και άλλους οι οποίοι είναι σε μια διαδικασία μαθητείας μέσα από το διαβίου μάθησης. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να, να αλλάξει η λέξη φοιτητέ πανεπιστημιακή δηλαδή, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί σαν έννοια η ιδέα ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι σε μαθητική διαδικασία, σπουδαστέ ή άλλοι, ε, καλύπτονται από το εράσμο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα και το δεύτερο ως ερώτηση. Ξέρουμε ότι η διευκόλυνση για δάνεια σπουδαστικά δεν έχει δώσει καλά αποτελέσματα. Προβλέπεται ωστόσο μέχρι το τέλος του 2019 ε, ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός για αυτό το δανεισμό που δεν απορροφάται όμως. Υπάρχει δυνατότητα, μια και ακόμη δεν ε, φαίνεται να έχει καλή απορροφητικότητα, ε, τα κονδύλια αυτά να μετατοπιστούν προς το Εράσμους. Και μήπως έχουμε την ευκαιρία μέσα από την έκθεση για την απαλλαγή να τοποθετηθούμε στο θέμα αυτό. Δεν ε, το γνωρίζω, το ρωτώ μόνο. Γιατί ξέρουμε ότι από την διευκόλυνση αυτή για το δάνειο υπάρχει η δυνατότητα να καταβάλλονται ποσά. Επομένως υπάρχει δυνατότητα της μετατόπισης, εν αναμονή ε, του να λειτουργήσει καλύτερα το σύστημα του δανεισμού αυτό. Δεν θα ήταν κρίμα να χαθούν τα χρήματα και τελικά να επανέλθουν στα Υπουργεία Οικονομικών των κρατών μελών. Θα ήταν πολύ μεγάλο κρίμα να χαθούν από τον τομέα το δικό μας. Το λέω απλά. Και τώρα παρακαλώ την Επιτροπή να λάβει το λόγο, εάν έχει την καλοσύνη. Παρακαλώ. Uh, to respond on the point about the... Θα ήθελα να πω ότι είμαι από την ε, Γενική Διεθνή και σε ό,τι αφορά το θέμα των ε, φοιτητών σπουδαστών σε κάθε δημοσιονομικό έτος προτείνουμε ανακατανομή των αδιάθετων κονδυλίων από τα επενδυτικά ταμεία για το μηχανισμό αυτό. Ήδη το έχουμε προβλέψει και το έχουμε προγραμματίσει. Ο κύριος Δρογεύσκη, για την τελευταία ερώτηση δεν είναι πια επίκαιρη γιατί απάντησε ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνήθως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά γρήγορα και μάλιστα και προληπτικά μερικές φορές προτείνει ανακατανομή των αδιάθετων κονδύλιων, οπότε δεν πάνε χαμένα. Σε ό,τι αφορά τώρα τον αριθμό των φοιτητών σπουδαστών, κύριε Πρόεδρε, δίκιο έχετε. Δεν είναι μόνο φοιτητέ, δεν είναι μόνο αθλητέ, αλλά είναι νέοι και λιγότερο νέοι και όλο και διευρύνεται το πρόγραμμα. Γι' αυτό έχει περιλάβει τώρα και το διδακτικό προσωπικό και δασκάλους καθηγητές, οπότε η ομάδα των δικαιούχων είναι όλο και μεγαλύτερη. Προσοχή λοιπόν, ο αριθμός των φοιτητών φάνηκε στους δείκτες της Επιτροπής ε, και στις κατευθυντήριες γραμμές που δώσαμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών από την ΚΟΥΛΤ. Και αυτό είναι ε, παράδειγμα μόνο, ε, γιατί δεν είναι μόνο οι φοιτητέ που συμμετέχουν στα προγράμματα του Erasmus Plus. Σε ό,τι αφορά τι προτάσει του κυρίου Μοργάνο, να γίνονται ταχύτερα οι δημοσιεύσεις. Πολύ εύστοχη αυτή η παρατήρηση. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι έχουμε ελάχιστο χρόνο ε, να εξοικειωθούμε με το θέμα και να εκδώσουμε τη γνωμοδότηση. Ενώ μετά είναι πολύ χρονοβόρη διαδικασία της ψηφοφορίας και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Θα ήταν πολύ καλύτερο να είχαμε τουλάχιστον δύο εβδομάδες περισσότερο για την εξέταση. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια της κυρίας Χέλγα Τρίπελ. Ε, επαναλαμβανόμαστε γιατί τακτικά και επανειλημμένως μιλούμε για την ελληπή χρηματοδότηση δύο προγραμμάτων και ζητούμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε αυτά τα δύο προγράμματα. Ε, και υπάρχουν πολλές θετικέ αξιολογήσεις ε, σχεδίων που δεν φτάνουν στο επίπεδο τη χρηματοδότηση γιατί δεν υπάρχουν ε, αρκετά μέσα. Και πάντως, αν συγκρίνουμε τους δείκτες απορρόφησης και εκτέλεση των δικών μας προγραμμάτων σχέση με άλλε επιτροπές, βρισκόμαστε χαμένοι γιατί έχουμε και λιγότερα μέσα και λιγότερα προγράμματα και δεν γίνονται αρκετές διορθώσεις. Και επίσης δείκτες 15-18% ε, είναι από τους χαμηλότερους δείκτες από όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε είναι κάτι που επαναλημμένως το επισημαίνουμε. Και για να αποφευθούν οι παρεξηγήσεις θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις μας και κάνει κάποιες διορθώσεις. Επαναλαμβάνω όμως ότι οι διορθώσεις είναι ανεπαρκείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απορρίπτει τη γνωμοδότησή μας, αλλά δεν ε, μας ικανοποιεί επαρκώς. Δεν λαμβάνει πλήρως υπόψη τις συστάσεις μας. Ευχαριστώ. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Υπενθυμίζω, προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών 16 ενδεκάτου στις 12. Και μετά θα υπάρχει βέβαια χρόνος για να συζητηθούν κάποια πράγματα στις συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών και ίσως να δοθούν και πιο συγκεκριμένες μορφές. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία στην περαιτέρω εργασία σας. Προχωρώ στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως που είναι η εξέταση σχεδίου γνωμοδοτήσεως για την δημιουργία του μέσου γειτονία για την αναπτυξιακή συνεργασία και τη διεθνή συνεργασία με εισηγήτρια την Μαρή Τερέζ Χιμένες Παμπάρ και προθεσμία καταθέσεων τροπολογιών 14 ενδεκάτου στις 2 το απόγευμα. Στις 22 Ιανουαρίου θα γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή Πολιτισμού. Οι δε αρμόδιες επί της ΑΦΕΤ και ΝΤΕΒΕ θα ψηφίσουν στις 4 Φεβρουαρίου. Να δώσω το λόγο αμέσως στην κυρία Χιμένες Μπαμπάτς. Κάπου την είδα προηγουμένως. Α, σας βλέπω, ναι. Ορίστε παρακαλώ. Μαρίτερε, έχετε το λόγο. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Η γνωμοδότησή μας αντρυπεί ε, στο θέμα της ε, επιρροής που έχει ο πολιτισμός στις ε, εξωτερικές σχέσεις και κυρίως στις πολιτικές ανάπτυξη και διεθνούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 89,2 δις είναι ο προπολογισμό αυτού του μηχανισμού και έχει τρεις πυλώνες, ένα γεωγραφικό, ένα θεματικό και ο τρίτος πυλώνας είναι η άμεση ταχεία αντίδραση. Στη συζητήση που έγινε σε επιτροπέ ΑΦΕΤ και ΑΝΤΕΒΕ, που είναι καθήλια αρμόδιε για την έκθεση αυτή, αμφισβητήθηκε ε, η νομοποίηση αυτού του μηχανισμού που θέλει να πλουστεύσει και να κάνει πιο ελαστικά τα χρηματοδοτικά μέσα της εξωτερικής πολιτικής. Σίγουρα είναι ανεπαρκή η αρχιτεκτονική αυτών των μέσων και είναι ανελαστικά σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα να ανταποκριθούν άμεσα στι αναδυόμενε προκλήσει. Γι' αυτό θεωρώ ότι χρειάζεται νέα αναθεώρηση για να αρθούν τα νομικά κολλήματα και τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Βέβαια, η νέα δομή δεν θα πρέπει να επηρεάσει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον προγραμματισμό και την εφαρμογή του νέου μηχανισμού και στην ελεκτική διαδικασία αυτού του μηχανισμού. Σε ό,τι αφορά τι δικέ μα δράσει, ο κανονισμό προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ελάχιστου στόχου και ήταν ελάχιστα φιλόδοξη κατά τη γνώμη μας η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Θα πρέπει να προβάλλουμε περισσότερο και να αναδείξουμε την παιδεία και τον πολιτισμό σε εξωτερικές σχέσεις και στην εξωτερική συνεργασία, διεθνή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτείνουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή ο μηχανισμό χρηματοδοτεί δράσει κινητικότητα μεταξύ των χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτε χώρε, αποκλειστικά μέσω του προγράμματο Έρασμο. Εμεί προτείνουμε να συμπεριληφθεί και το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη έτσι θα αναδείξουμε το ρόλο του πολιτισμού και των δημιουργικών επιχειρήσεων στις εξωτερικές αίσθησει τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα μπορούμε να προωθήσουμε την κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη και τον διαπολιτισμικό διάλογο. Δεύτερον, θα πρέπει να εξάρουμε το ρόλο που έχει η παιδεία χωρίς αποκλεισμούς και η ποιοτική παιδεία για να μειωθεί η φτώχεια και οι ανισότητες. Ε, να ενισχυθεί η ανοχή, να καταπολεμηθεί η μισελοδοξία και να διαμορφώσουμε πιο ειρηνικέ κοινωνίε. Άλλωστε η παιδεία είναι ο στόχο 4 του θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, ε, ε, έχουμε και ένα φιλόδοξο αίτημα. Προκειμένου να προωθήσουμε τη διεθνή διάσταση τη παιδεία και του πολιτισμού, ζητούμε να αφιερωθεί τουλάχιστον 15% του πολιτισμού στι δράσει παιδεία και πολιτισμού. Αξιότιμοι συνάδελφοι, δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε πόσο σημαντικό είναι ο πολιτισμό και η παιδεία στι εξωτερικέ μα σχέσει και στι πολιτικέ μα για τη διεθνή συνεργασία. Δυστυχώ όμω πρέπει να κάνουμε αυτή την επανάληψη και μάλιστα σύσσωμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και στη συνεργασία με τους συναδέλφους μας σε επιτροπές ΑΦΕΤ και ΔΕΒΕ. Είμαι στη διάθεσή σας για να συζητήσω τις προτάσεις ε, και τις παρατηρήσεις σας. Σα ευχαριστώ για την προσοχή. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ευχαριστώ πολύ, Μαρή Τερέζ. Οι σκιώδεις ηγητές ακολουθούν τώρα και πρώτος ο κύριος Στογεύσκη. Θα ήθελα καταρχήν να επισημάνω ότι σε 23 μήνες θα εκπνεύσει αυτό το πρόγραμμα, οπότε έχουμε πολύ μικρή προοπτική σε ό,τι αφορά την υλοποίησή του. Δεύτερον, ε, ως Επιτροπή Πολιτισμού δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο μας γιατί ζητούμε τα προγράμματα μας όπως Δημιουργική Ευρώπη, Ευρώπη των Πολιτών και Ορίζοντας 2020 ε, και ο συνδυασμό τους ε, ίσως ε, οδηγεί σε περικοπή του προϋπολογισμού των προγραμμάτων ενώ έχουμε επιπλέον προκλήσει τα πλαίσια του προγράμματος που ούτως ή άλλως έχει 90 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί στις παρατηρήσεις μας γιατί αν θέλουμε να συνδέσουμε διάφορα προγράμματα που ούτω ή άλλω υποχρηματοδοτούνται, όπω έχουμε πει, και αν θέλουμε να τα συνδυάσουμε και με άλλε για να καλύψουν και άλλε επιπλέον δράσει, αυτό θα είναι υπερβολικό. Πάντω, δίκιο έχει συνάδελφο ότι το θέμα του πολιτισμού και τη παιδεία θα πρέπει να αξιοποιηθούν ω μέσα για να ε, βελτιωθούν τα σημεία που είναι τα πιο σημαντικά στη, την πολιτική γειτονία και την πολιτικού διεθνού συνεργασία. Οπότε, οι δύο συνιστώσει, η γεωγραφική και η θεματική, μπορούν να συμπληρωθούν με τις τροπολογίες μας. Σε ό,τι αφορά και τη συνιστώσα τη ταχεία αντίδραση, ουδέποτε δεν λαμβάνονται υπόψη ο πολιτισμός και η παιδεία ω στοιχεία που μπορούν να βελτιώσουν την ταχεία μα αντίδραση. Οπότε θα πρέπει να φροντίσουμε κυρίως δύο στοιχεία στη γνωμοδότησή μας. Καταρχήν, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τον πολιτισμό, την παιδεία και τα άλλα θέματα των αρμοδιοτήτων μα, χωρί όμω ε, να μειώνουμε ή να επηρεάζουμε αρνητικά οικονομικά τα προγράμματα. Επίσης, με τις τροπολογίες μας θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στα πλαίσια των εργαλείων και του το μηχανισμού ε, της ε, πολιτικής, της εξωτερικής πολιτικής και της γειτονίας, ο πολιτισμός και η παιδεία μπορούν να διδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τζούλι Ward. Ευχαριστώ, αγαπητή Πρόεδρε, και ευχαριστώ την κυρία Χιμένες Παρμπάτ για την δουλειά που έκανε και το θαυμάσιο σχέδιο που μας υποβάλλει. Οι τροπολογίες που προτείνει αποδίδουν τη μεγάλη σημασία και οριζόντια σημασία της πολιτισμικής παιδείας για εξωτερικές δράσεις της Ένωσης, συνεργασία με γειτονικέ χώρες και πολιτικές αναπτύξεις. Θα τονίσω ορισμένα από τα πράγματα που με ενδιαφέρουν ιδιαίτερος και την ομάδα μου. Ανάγκη προώθησης δηλαδή των διαπροσωπικών επαφών και πολιτισμικών για την επιτεύξη των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, για την πρόσβαση στην εκπαίδευση ως ε, ανθρώπινο δικαίωμα και για το τελευταίο αυτό θέμα θα ήθελα, έχουμε καταθέσει τροπολογία, για να δημιουργηθούν εκπαιδευτικοί διάδρομοι για νέους και παιδιά σε ζώνες συγκρούσεων. Τροπολογίες θα καταθέσω επίσης για την ανάγκη περαιτέρω πρόθεση της κοινωνίας των πολιτών και τη στήριξη των φορέων της. Αυτά για τις ε, καθεαυτές αρμοδιότητες της ε, Επιτροπής μας. Κάτι με ανησυχεί όμως την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με την προτινόμενη νομική βάση βλέπω μία τάση να συνδέσουν στόχους πολιτικής της ανάπτυξης με τις αιτίε της μετανάστευσης. Ναι, η αναπτυξιακή συνεργασία μπορεί να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την ευμερία ατόμων και κοινοτήτων, να αντιμετωπιστούν κάποιες αιτίε ε, μετανάστευσης, αλλά δεν μπορούμε να μειώσουμε τον χαρακτήρα αυτού του κρίσιμου εργαλείου μόνο στην προσπάθεια επίτευξης αυτού του στόχου, ξεχνώντας τις βασικές αξίες της ανάπτυξης και της συνεργασίας. Και μιλώ ως ε, ένα πρόσωπο το οποίο έχει πάρει και μάστερς για θέματα ανάπτυξης, από το πανεπιστήμιο δηλαδή. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικές και προσεκτικοί όταν ε, ανακατεύουμε μετανάστευση και ανάπτυξη. Σας ευχαριστούμε. Jill Evans. Ορίστε Jill. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη γνωμοδότησή της που νομίζω ότι τονίζει ακριβώς την ανάγκη αναφοράς σε πολιτισμό και εκπαίδευση στο σχέδιο κανονισμού. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συνδυαστούν πολιτικές δημιουργίες της ειρήνης, ανάμυνας και μετανάστευσης είναι με ε, ε, μια πρόσβαση, αλλά πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά ωστόσο τον πολιτισμό, οι διεθνείς επαφές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών χρειάζονται και ισχυρές πολιτισμικές διασυνδέσεις για να επιτύχουν. Ο διάλογος είναι ουσιώδης για να επιτευθεί μια πλέον ειρηνική ε, σχέση και να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε κοινέ αξίες και να εξεύουμε κοινέ ευκαιρίες. Όπως λέχθηκε ήδη η Δημιουργική Ευρώπη, ο Έρασμος και άλλα ε, σχετικά προγράμματα θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων. Να δώσουμε λοιπόν προτεραιότητα στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος σε κρίσεις, σειράξεις, συγκρούσεις και αυτά να τα βάλουμε, μάλλον τον πολιτισμό να τον βάλουμε στην καρδιά των προσπαθειών μας. Υποστηρίζουμε την γραμμή που ακολουθεί η εισηγήτρια στην ομοδότησή της. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τρίπελ στα αγγλικά. Ευχαριστώ. Μετά τα όσα είπε η φίλη μου Τζιλ, θέλω να τονίσω και εγώ πόσο σημαντικό είναι στις ε, εξωτερικές μας σχέσεις να περιλαμβάνουμε παιδεία, πολιτισμό και αλλαγή του κλίματος. Έχω και μια εμπειρία. Μόλις επιστρέφω από το Μπάλι, όπου διεξήχθη διάσκεψη σκηνοθετών, ε, συγγραφέων, ακτιβιστών και άλλων που ασχολούνται με τη βιωσιμότητα για όλα αυτά τα πλαστικά σκουπίδια και αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο ε, αλλαγής κλίματος και της αύξησης του επίπεδου των νερών που απειλεί τα νησιά αυτά. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το συνέδριο αυτό, διότι αναφέρθηκε στο τι μπορούν να κάνουν οι συγγραφείς, ακόμα και με ποίηματα και τέτοια, και για όλα αυτά τα θέματα της βιωσιμότητας, για την προστασία των ωκεανών, πώς μπορούν να καθαρίσουν τα νερά και πώς μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά τα οικολογικά, μαζί με τα θέματα των μεταφορών, ώστε οι μεταφορές να γίνουν δέτερες σε ό,τι αφορά τις εκπομπές και αυτά να συνδυαστούν με τις αφηγήσει, διηγήσει, ε, παραδόσεις των διαφόρων λαών. Οι άνθρωποι όταν συνέρχονται μπορούν να συζητήσουν και να πούν τέτοια πράγματα. Υπήρχε κάποιο από το Μιανμάρ, από την Νότια Αφρική, από τι Ηνωμένε Πολιτείε, βέβαια από το Μπαλί, από την Ινδονησία, Γερμανοί. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι είναι καλό να διατηρούμε επαφές με τους ανθρώπους που οργανώνουν τέτοια συνέδρια που θα έπρεπε να εντάσσονται στο πρόγραμμά μας. Αν συνδυάσουμε τις ιδέες μας με τις δικές τους, νομίζω ότι μπορούμε να ασκήσουμε πολύ μεγαλύτερη επιρροή. Το πάλι βεβαίω είναι μόνο ένα παράδειγμα. Υπάρχουν και άλλες σχετικές ιδέες και πρωτοβουλίες που αναφέρονται βέβαια στην συνεργασία και στις επαφές. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως θέλει να λάβει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ορίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σας. Ναι, όντως, μπορώ να πω δύο λόγια, καλώς ορίζοντας την έκθεση. Συμφωνούμε με το Κοινοβούλιο πως χρειάζεται περισσότερη ευελιξία για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων μας στην εξωτερική δράση. Πρέπει να υπογραμμιστεί η σημασία της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, τομείς που σαφώς αναφέρονται και στους στόχους της ε, βιώσιμης ανάπτυξης και άρα προβλέπονται και τα σχετικά εργαλεία γιατί η κατάλληλη εκπαίδευση είναι ένα ε, όπλο με το οποίο μπορούμε να πολεμήσουμε την φτώχεια και μπορεί να στήριξει την ανάπτυξη του ανθρώπου. Μέσα σε αυτό βέβαια εντάσσεται και ο πολιτισμός. Έτσι λοιπόν οι προτάσεις είναι ευπρόσδεκτες με μόνο ζήτημα τον προσδιορισμό πολλών και συγκεκριμένων στόχων στο κείμενο. Με 15% στόχο για την εκπαίδευση και την, τον πολιτισμό που έρχεται αντίθετο, σε αντίθεση με την αρχή της ε, ιδιοποίησης. Και της προτίμησης για το πρόγραμμα που είναι ένα κομμάτι του εργαλείου. Προσπαθούμε λοιπόν ε, όταν αναπτύσσουμε συνεργασία με χώρες εταίρους να την αναπτύσσουμε από κοινού μαζί με τους άλλους χορηγούς αλλά δεν θέλουμε να περιπλέξουμε τα πράγματα σχέση με το πώς θα υλοποιηθούν όλα αυτά. υποστήριξη στον πολιτισμό και την εκπαίδευση καλύπτεται στα παραρτήματα και στον τομέα ε, γεωγραφική συνεργασία ως στόχο, αλλά και στο θεματικό πρόγραμμα που συμπληρώνει τα γεωγραφικά. Τα αναγνωρίζει λοιπόν το μέσον. Στη δημιουργική Ευρώπη επίσης, που δεν αναφέρεται ρητά το μέσον αυτό. Ωστόσο προβλέπεται η δυνατότητα για τη χρηματοδότηση μέσω της Δημιουργικής Ευρώπης ε, και συνεργασιών με τις χώρες εταίρους ανά τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεση λοιπόν και βεβαίως θα συνεχιστούν οι συνομιλίες ε, για το θέμα αυτό. Vielen herzlichen Dank, παρακαλώ. Καταλαβαίνω απόλυτα το φόβο που έχουμε να απογυμνώσουμε έναν Άγιο για να ντύσουμε άλλο. Δηλαδή να αφαιρέσουμε κονδύλια από ένα πρόγραμμα για να χρηματοδοτήσουμε άλλο. Να βγάζουμε από τη μία τσέπη και να βάζουμε στην άλλη. Ε, αυτό που θελήσαμε για το έρασμό είναι να μπορεί να χρηματοδοτεί και τη δημιουργική Ευρώπη. Ακριβώς για να προωθήσουμε τους στόχους μας. Δηλαδή να αντιμετωπίσουμε τον πολιτισμό με πιο ευρία έννοια. Αυτός ήταν ο στόχος όταν προτείναμε συνδυασμό. Και ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους, τις ιδέες και τα σχόλιά τους. Ε, οι συνεργάτες μου ε, είναι στη διάθεσή σας και εγώ είμαι πρόθυμη και οι πόρτες στο γραφείο μου ανοιχτέ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, 14 Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι προθεσμία, 22 Ιανουαρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. πολύ καλή δουλειά και πολύ καλές προσδοκίες για τα πολύ καλά αποτελέσματα από τη συνεργασία με τους Κιώδης. Σας ευχαριστώ πολύ και την κατάλληλη στιγμή ήρθε και η προσκεκλημένη για το επόμενο θέμα της ημερήσιας δάταξης. Προχώρησαμε λίγο ταχύτερα από ό,τι προσδοκούσαμε σήμερα. Χαίρομαι όμως που καταφέρατε να φτάσετε πιο νωρίς κι εσείς. Σημείο 7 στην ημερήσια διάταξη. Καλώς ορίζω πρώτα τον προσκεκλημένο μας. Nein, das, äh, das ist immer so. so. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Μελέτη που έχουμε αναθέσει στο Policy Department για τον τομέα των οπτικοακουστικών και τις συνέπειες σε αυτόν του Brexit. Έχουμε τον Μαρκόλ, ε, εμπειρογνώμονά μας από το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού Δικαίου των ΜΜΕ. Τον Απρίλιο του 2017 ξεκίνησε αυτή η μελέτη και Βλέπουμε ότι και από τις δικές μας εκθέσεις βεβαίως ότι μέχρι τώρα η διαδικασία του Brexit δεν έχει φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχέση με τη διαμόρφωση των των οπτικοακουστικών αλλά και άλλων ε, τομέων. Παραμένει λοιπόν να σε αφήσει η κατάσταση, αλλά το μέσο των οπτικοακουστικών έχει πολύ μεγάλη σημασία και καθώς όλα αυτά παραμένουν σε μια αχλή, είμαστε υποχρεωμένοι να επεξεργαστούμε διαφορετικά σενάρια και εναλλακτικέ εξελίξεις για το μέλλον και να προετοιμαστούμε αναλόγως. Ε, όπως είπαμε, χαρά, καλώ ορίζω εδώ τον Μαρκ Κόλ, τον ε, εκπρόσωπο, τον απεσταλμένο από, την, ε, από τον τομέα των οπτικοακουστικών, του οπτικοακουστικού δικαίου του Πανεπιστημίου του Λουξεμβούργου και περιμένουμε να ακούσουμε τι βλέπετε για το μέλλον του Brexit στον τομέα των οπτικοακουστικών. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο και χαίρομαι που σας βλέπω εδώ. Πριν περάσω στα γερμανικά, σας ευχαριστώ και εγώ κυρία Πρόεδρε για τη δυνατότητα που μου δίνετε σήμερα να κάνω την παρουσίαση σήμερα. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού, Χάρηκα ιδιαίτερω όχι μόνο γιατί εκπώνησα τη μελέτη, αλλά και μου δίνεται ευκαιρία να σα παρουσιάσω τα βασικά τη πορίσματα. Σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο, βέβαια, όπω θα φαντάζεστε, θα είναι αδύνατο να σα παρουσιάσω ολόκληρη τη μελέτη. Θα σταθώ σε μερικά μόνο σημεία. Πάντω, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι τρει είναι οι βασικέ διαστάσει, ή μάλλον δύο. η οδηγία για την υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων και οι συνέπειε τη και ε, πώς θα εφαρμοστούν τα πνευματικά δικαιώματα στον οπτικοακουστικό κλάδο και τι ρόλο θα διαδραματίσουν. Θα ήθελα καταρχήν εν συντομία να σας παρουσιάσω γιατί είναι τόσο σημαντικό το Brexit και ότι θα έχει σημαντικές συνέπειες για τον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων. Τα οπτικοακουστικά μέσα είναι μη διάσουσα πτυχή που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στο Brexit και όπως είπε η Πρόεδρος δεν ξέρουμε πώς θα δρομολογηθεί και τι μορφή θα λάβει το Brexit. Οπότε θα πρέπει να ε, ε, να εξερευνήσουμε διάφορα σενάρια ανάλογα και με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Θα σα κάνω μια παρουσίαση και αν υπάρχουν απορίε θα επανέλθουμε σε επιμέρου θέματα. Καταρχήν, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι παρόλο που είναι θέμα κοινή λογική, θα πρέπει να επισημάνουμε πόσο ε, σημαντικέ είναι οι εξελίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα οπτικοακουστικά μέσα. Τα τελευταία 30 χρόνια είχαμε μια σειρά κανονισμών και οδηγιών που συνδέθηκαν μεταξύ τους και διαμόρφωσαν όλο το περιβάλλον των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ε, προκειμένου να αναπτυχθεί η διασυνοριακή πρόσβαση και η διάδοση περιεχομένου. Χωρίς το ενωσιακό δίκαιο δεν θα είχαμε τη σημερινή αγορά οπτικοακουστικών μέσων, υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων. Και τώρα, τι μας ενδιαφέρει εδώ το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, θα γνωρίζετε όλοι ότι όχι μόνο ποσοτικά το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το σημαντικότερο κόμβο των παρόχων οπτικοακουστικών υπηρεσιών, αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό ότι πολλοί πάροχοι που ε, βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, απευθύνονται προς άλλους προορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι αποκλειστικά μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και ακόμη με την πολιτισμική πολυμορφία εντό των κρατών μελών και εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε ένα είδο Ευρωπαϊκή Αγορά που διαφέρει κάπω από την βορειοαμερικανική αγορά οπτικοακουστικών μέσων. Και εδώ τα κοινά σημεία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ περισσότερα από τι διαφορέ. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό τι είδου Brexit τελικά θα έχουμε. Γιατί από αυτό θα εξαρτηθεί και το πόσο σκληρό ή επιθένει το Brexit ε, θα επηρεαστεί ανάλογα ο κλάδος των οπτικοακουστικών μέσων. Ε, μην φοβάστε με τη διαφάνεια που θα σας δείξω, που αφορά το πρώτο κεφάλαιο της μελέτης. Καταρχήν, ξεκινώντας από τα αριστερά προς τα δεξιά, ε, η αριστερή πλευρά δείχνει τη μεγαλύτερη δυνατή σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η δεξιά πλευρά είναι αν δεν έχουμε τίποτα, καμία συμφωνία. Και τίποτα δεν σημαίνει φυσικά το απόλυτο μηδέν αλλά σίγουρα το καλύτερο θα ήταν να συνεχιστεί η αγορά με τη μορφή που έχει τώρα, με στενή συνεργασία δηλαδή, στα πλαίσια τη συμμετοχή στον ΕΟΧ, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Και στα πλαίσια του ΕΟΧ έχουμε ελάχιστε διαφορέ σε σχέση με το δικό μα οπτικοακουστικό κλάδο. Ε, Ανάλογα με το αν είναι κανεί πλήρε μέρο Ευρωπαϊκή Ένωση, αν εφαρμόζει την ομοθεσία με βάση τι αρχέ του ΕΟΧ γιατί έχουμε ουσιαστικά το ενωσιακό δίκαιο που εφαρμόζεται στο νέο. Ακόμη και η παρακολούθηση και η υποπτία της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου είναι η ίδια με το ΝΕΟΧ. Τώρα, άλλο σενάριο είναι το νορβηγικό μοντέλο, όπως λέμε. Ε, και ένα νομικά ενδιαφέρον ζήτημα επίσης, αλλά μάλλον πολιτικά απίθανο να ε, διαφυσβητηθεί, είναι αν θα μπορούσε το, το Ηνωμένο Βασίλειο να γίνει αυτόματα μέλος του ΕΟΧΑ, μια και έχει υπογράψει τη συμφωνία του ΕΟΧΑ ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παραμείνει μέλος του ΕΟΧ και μετά τον Brexit. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, μάλλον απίθανο είναι αυτό. Κανένας δεν θα ε, ρωτήσει αν ε, το Ενωμένο Βασίλειο παραμείνει μέλος του ΕΟΧ χωρίς να το ζητήσει συγκεκριμένα. Πάντως, αν μείνει στον ΕΟΧ, θα, θα διατηρηθεί η συνεργασία στον ίδιο βαθμό όπως και σήμερα. Δεύτερο σενάριο είναι ΕΖΕΣ, η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ή επιπλέον διμερή συμφωνία. Εδώ θα είχαμε το ελβετικό μοντέλο. Αλλά ούτε και για αυτό το θέμα ε, ε, εξέφρασε κάποια σχετική επιθυμία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, θα μπορούσαμε να έχουμε είτε μια τελωνιακή ένωση, είτε μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Σε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών όμω, θεωρητικά για τα οπτικοκοστικά μέσα θα λέγαμε εντάξει, κανένα πρόβλημα, θα συμπεριλάβουμε όλου του τομεί που έχουμε σήμερα και που καλύπτονται από την οδηγία για τι υπηρεσίε των οπτικοακουστικών μέσων. Βέβαια, αν αναλύσουμε τι ε, συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών στο παρελθόν, ουδέποτε δεν κάλυπταν αυτέ και τον τομέα οπτικοακουστικών μέσων. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μία ε, πολιτιστική εξαίρεση. De facto δηλαδή ουσιαστικά οι υπηρεσίε οπτικοακουστικών μέσων ε, εξαιρούνται από τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και υπάρχουν εύλογοι λόγοι γι' αυτό. Γιατί σε μια κανονική συμφωνία FTA αποκλείεται να έχουμε ξαφνικά επέκταση και στα οπτικοακουστικά μέσα. Ισχύει η πολιτιστική εξαίρεση. Τώρα, τι γίνει αν δεν έχουμε καμία συμφωνία, αν δεν έχουμε λεπτομέρεια ειδικούς ε, κανόνες για τα οπτικοακουστικά μέσα. Αυτό το τίποτα που λέμε εντός εισαγωγικών. Οπότε θα εξακολουθούν να ισχύουν οι κανόνες του παγκόσμ... της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Και το Ηνωμένο Βασίλειο ήδη έχει ε, κυρώσει πολλές συμφωνίες στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ε, για την διασυνοριακή τηλεόραση, για παράδειγμα, έχει υπογραφεί η σχετική συμφωνία, η σύμβαση που αναπτύχθηκε εκ παραλίλου με την οδηγία για τηλεόραση χωρίς σύνορα, που ήταν ε, προ πρόδρομος της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Βέβαια, ίσως δημιουργηθούν κάποια κενά και υπάρχουν προβλήματα, γιατί δεν έχουν κυρώσει όλα τα κράτη-μέλη τη σύμβαση αυτή, οπότε και εκεί θα υπάρξει διαφορά στη σχέση μεταξύ κάποιων κρατών μελών με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και υπάρχει και η σύμβαση για την διασυνοριακή τηλεόραση, που έχει κολλήσει ουσιαστικά στην κατάσταση των τελών της δεκαετίας του 90. Δεν έχει γίνει επικαιροποίηση και ενημέρωση ώστε να λαμβάνεται υπόψη η νέα έννοια των ΜΜΕ, όπως αναφέρεται στην οδηγία της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων. Οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν θα έχουμε μάλλον αντικατάσταση. Σε ό,τι αφορά τα GATS, και εκεί έχουμε τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που καλύπτονται καταρχήν, αλλά τα κράτη-μέλη του GATS δεν έχουν δεσμευτεί για συγκεκριμένα θέματα του τομέα. Οπότε, αν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του ΓΚΑΤΣ, την χάνουν καλύτερη μεταχείρισης, μπορούν να το κάνουν. Αλλά αν το Ηνωμένο Βασίλειο βρεθεί εκτός ενιαίας αγοράς, δεν θα λάβει αυτή την προτιμησιακή μεταχείριση. Γιατί αν το κάνουν αυτό για το Ηνωμένο Βασίλειο, το θέμα τη προτιμησιακή μεταχείριση στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να το επεκτείνουν και σε άλλε χώρε του κόσμου. Κάτι που δεν θα το θέλουν. Τώρα, τι γίνεται με την οδηγία AVMSD, την οδηγία για τι υπηρεσίε οπτικοακουστικών μέσων. Ε, Προχθέ ε, έχει ληφθεί μια συμφωνία και η βασική αρχή είναι η χώρα προέλευση, η αρχή τη χώρα προέλευση, που διαμόρφωσε μια ευρωπαϊκή αγορά που οι πάροχοι πια μπορούν να επιλέξουν τον τόπο κατάστασή τους και να μπορούν ε, να εκπέμπουν παντού στην Ευρώπη. Οπότε έχουμε ένα είδος ε, one-stop shop, μόνο ενιαία θηρίδας, η μονοπευθυντική θηρίδας. Και μερικές φορές αναφέρεται, δεν έχουμε μια εφαρμογή της πλήρους αρχής ε, Τη χώρας προέλευση γιατί υπάρχουν εξαιρέσει και διαδικασίε που προβλέπουμε, αλλά επαναλαμβάνω είναι ε, ε, και δεν ε, αποδυναμώνουν την αρχή τη χώρα προέλευση. Απλώ υπάρχουν κάποιες παρεκκλήσεις εξαιρέσει Καταρχήν να, να προσδιορίσουμε ποια είναι η χώρα προέλευση και ποια δικαιοδοσία ισχύει. Γιατί αυτή τη στιγμή η δικαιοδοσία για πολλούς ε, παρόχους είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί εκεί έχουν την έδρα τους εκεί έχουν τον τόπο εγκατάσταση. Πάντως, η οδηγία έχει και ένα επικουρικό κριτήριο που λέει ακόμη και αν δεν υπάρχει έδρα εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον για τους παρόχου που χρησιμοποιούν ε, δορυφορικέ υπηρεσίες ή ε, uplink προς ε, δορυφορικές υπηρεσίες, υπάρχει δυνατότητα να θεωρηθούν ότι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στη δικαιοδοσία κάποιας χώρας μέλους. Τώρα, αν στηριχθούμε μόνο σε αυτό το επικουρικό κριτήριο για τον πάροχο, αυτό δεν είναι και πολύ ασφαλές. Γιατί τι θα πει, αν έχει κάποιο τόπο εγκατάσταση ή ένα παράρτημα ή τα κεντρικά γραφεία, είναι εύκολο να δούμε τη δικαιοδοσία, αλλά σε τέτοια περίπτωση δεν θα είναι εύκολο να την διαπιστώσουμε. Άλλο θέμα, το θέμα των ποσοστώσεων στην οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Και ένα μεγάλο τμήμα του περιεχομένου που θεωρείται ευρωπαϊκό έργο παράγεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι από του σημαντικότερου παραγωγού περιεχομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα τι θα γίνει, θα καταργηθούν οι ποσοστώσει, όχι, γιατί στην οδηγία για, τα, για τι υπηρεσίε των επιτικοπιστικών μέσων τα ευρωπαϊκά έργα είναι έργα που ε, γίνονται από εταίρου που έχουν υπογράψει τι συμβάσει του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Κάτι που ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε ε, τα έργα που παράγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ε, ε, θεωρούνται και πάλι ευρωπαϊκά για το δικαστήριο. Πάντως, στην οδηγία προβλέπεται αυστηρή υποχρέωση υποβολής εκθέσεων. Ε, μετά τον Brexit όμως και χωρίς συμφωνία δεν θα υποχρεούται για να υποβάλει δηλώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε θα είναι ε, δύσκολο να δούμε αν τα η, προ, η προέλευση των έργων είναι όντως το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί δεν θα υπάρχει πλέον υποχρέωση υποβολής εκθέσεων οπότε θα, μπορέσω, θα είναι δυνατόν να έχουμε κάποια έργα που θα παράγονται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου θα χαρακτηρίζονται έργα του Ηνωμένου Βασιλείου και αυτό θα είναι δύσκολο να το εξακριβώσει το δικαστήριο χωρίς την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων. Και άλλο πρόβλημα με την οδηγία αυτή είναι η αναθεώρηση που αναμένεται φέτο, που θα είναι σημαντικό, μια σημαντική καινοτομία που θα ισχύει για τι πλατφόρμε κοινή χρήση βίντεο. Τώρα, μετά τον Brexit, αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν εφαρμόσει αντίστοιχου κανόνε στο εθνικό του δίκαιο, δεν υποχρεούται. Ε, ίσως θα είναι πιο ελκυστικό το Ηνωμένο Βασίλειο για πλατφόρμε κοινή χρήση βίντεο να βρίσκονται εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάνε δηλαδή στο Ηνωμένο Βασίλειο και να στοχεύουν προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντω, η νομοθεσία εδώ είναι αρκετά διορατική και υπάρχει δικαιοδοσία που λέει δεν είναι η βασική χώρα της, α, ε, ε, της αρχής χώρας προέλευσης και ακόμη και δεν υπάρχει κατάσταση σε μια χώρα, αν υπάρχει κάποια σχέση και αυτό ισχύει για τις πλατφόρμες κοινής χρήσης βίντεο, αυτός ο σύνδεσμος μπορεί να είναι αρκετός ώστε να θεωρηθεί ότι μια πλατφόρμα υπόκειται στη δικαιοδοσία αυτής της χώρας. Τώρα, Μία πλατφόρμα κοινή χρήση βίντεο κατά πάσα πιθανότητα θα εφαρμόσει του κανόνε ε, με τρόπο ώστε να μην ε, λαμβάνει υπόψη αν προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο ή από άλλη χώρα. Θα ε, θεωρήσουν οι πλατφόρμες την Ευρωπαϊκή Ένωση ω σύνολο, προκειμένου να τηρηθούν οι κατευθυντήριε γραμμέ τη οδηγία. Δεν θα πούν δηλαδή οι πλατφόρμε στοχεύουν προ την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτό. Και κάτι αντίστοιχο έγινε με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων και για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας μετά το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και από πλατφόρμες κοινή χρήση δεδομένων. Σε ό,τι αφορά την αγορά πνευματικών δικαιωμάτων, που είναι κάπως πιο περίπλοκη, γιατί για τα πνευματικά δικαιώματα, το copyright, υπάρχει υψηλό βαθμός εναρμόνισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μερικέ φορέ υπάρχει η λαθασμένη αντίληψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε αυτό που συμφώνησε ο Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματική Ιδιοκτησία με τον ΠΟΕ. Δεν ισχύει όμω κάτι τέτοιο. Το επίπεδο εναρμόνιση εντό Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ υψηλότερο. Ακόμη και ε, απέρευσε από τις διεθνείς συνθήκες. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ερμήνευσε τις οδηγίες με τέτοιο τρόπο που όχι μόνο ξεπερνά το στενό τους περιεχόμενο, αλλά έχει δώσει και πολλές κατευθυντήρες γραμμές στο δικαστήριο για, την εφαρμογή των οδηγιών. Οπότε ακόμη και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεσμεύεται από την ερμηνεία του δικαστηρίου. Και α, δεν, δεν, θα, μάλλον, δεν θα δεσμεύεται στο μέλλον από την ερμηνεία του δικαστηρίου. Οπότε οι ερμηνείες για τα copyright θα είναι διαφορετικές σε περίπτωση που το Brexit ε, λάβει χώρα χωρίς συμφωνία. Επίσης, στα πλαίσια των διεθνών συμφωνιών που θα εξακολουθούν να ισχύουν μόνο αν παραμείνει κανεί μέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξασφαλίσει για του δημιουργού του την υψηλή προστασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αν έχουμε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών χωρί ειδικέ προβλέψει για τα οπτικοακουστικά μέσα, η πιθανότητα τη ε, διασυνοριακή διάδοση με την ίδια προστασία πνευματική ιδιοκτησία είναι μάλλον απίθανη. Και αν θέλουμε μια ειδική διάταξη που θα έχει το ίδιο επίπεδο προστασία με αυτό που ισχύει σήμερα, μάλλον θα είναι αδύνατο. Γιατί θα σας δώσω δύο παράδειγμα. Καταρχήν, αρχή ανάλωσης δικαιωμάτων, υποχρεωτικές ε, ε, διοδοτήσεις, εφορητότητα των δικαιωμάτων, εκαθάριση δικαιωμάτων δημιουργού, οι οδηγίες ATCAP και οι πιθανές προσθήκες. Για όλα αυτά τα θέματα, αν θέλουμε να τα συμπεριλάβουμε σε μεμονωμένη διμερή συμφωνία, αυτό θα είναι πολύ δύσκολο, γιατί μιλάμε για ένα πλέγμα κανόνων που θα διακυβευθούν μετά τον Brexit. Ποιες είναι λοιπόν οι βασικές μου παρατηρήσεις και έχω φτάσει στο τέταρτο που μου δώσατε. Πιστεύω το πλαίσιο τη οδηγία για τι υπηρεσίε οπτικοακουστικών μέσων είναι καλύτερα είναι εκτό παρά εκτό. Εντό παρά εκτό. Για να καλύπτονται όλοι οι πάροχοι. Είναι πολύ πιο δελαστικό για του παρόχου να καλύπτονται από την οδηγία EVMS παρά να εκπίπτουν. Γιατί υπάρχουν πολλέ υποχρεώσει με την οδηγία αυτή, αλλά σίγουρα τα ωφέλη από τη δυνατότητα εκπομπή σε όλη την Ευρώπη είναι πολύ πιο μεγάλα παρά να βρίσκονται εκτό δικαιοδοσίας Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή τη στιγμή έχουμε συζήτηση για την επέκταση των κανόνων στι πλατφόρμες. Και αυτή η συζήτηση είναι πολύ σημαντική και σίγουρα το Ηνωμένο Βασίλειο συνέβαλε σημαντικά στη συζήτηση αυτή. Αν τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο φύγει με σκληρό Brexit, αυτό δεν θα επηρεάσει τη συζήτηση στα θέματα αυτά, αλλά αν η Ευρωπαϊκή Ένωση χάσει το Ηνωμένο Βασίλειο από άποψη θεμελιωδών δικαιωμάτων για μια αγορά που έχουμε ελεύθερη διακίνηση της πληροφορίας και το περιεχομένου, αυτός δεν είναι επιθυμητός στόχος. Οπότε αν υπάρχει δυνατότητα να συμφωνήσουμε για στενή συνεργασία και συνέχιση των νομοθετικών διατάξεων και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό θα ήταν ευχής έργων. Χωρίς συμφωνία όμως θα δούμε πώς θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τη σύντομη αυτή ε, εντάχει επισκόπηση. Βλέπουμε βεβαίως ότι προβλήματα μπορεί να προκύψουν στον τομέα αυτών των οπτικοακουστικών από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μας περιμένει, πόσα εκρεμή μάλιστα ζητήματα παραμένουν ανεπίλητα ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν είναι δεδομένο ότι θα καλύψει όλα τα ζητήματα της μελλοντική συνεργασίας και έτσι είναι πολλά τα εκρεμή ζητήματα για τα οποία μόνο υποθέσεις μπορούμε να διατυπώσουμε. Αλλά είναι σημαντικό. Εκθέσαμε τα κύρια σενάρια και τις προτάσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που να προκύψουν από τη την άλλη εκδοχή. Θα παρακαλέσω τώρα τον κύριο Στρογεύσκη, που είναι και πρόεδρος της ομάδας εργασίας του Brexit, της Επιτροπής μας, να λάβει το λόγο πρώτος. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην ε, Επιτροπή για το Brexit ε, ήδη θέσαμε όλα αυτά τα ζητήματα που μας παρουσίασε ο κ. Καθηγητής και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτή την ε, συνοπτική αλλά μεστή παρουσίαση ε, που μας κρούσε το κόδωνα του κινδύνου γιατί αν δεν υπάρχει νομική λύση θα βρεθούμε σε ένα νομικό κενό που θα είναι πολύ επιζήμιο και για τις οπτικοακουστικές, ε, για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, αλλά και για τα δικαιώματα του δημιουργού και την πνευματική ιδιοκτησία, που ήδη είναι θέμα ε, που μας δημιουργεί προβλήματα. Ακούσαμε τις στάσεις σας και τα σενάρια, το νορβηγικό, το ελβετικό, το καναδέζικο μοντέλο, το τουρκικό μοντέλο. Θα μπορούσατε να μας ε, παρουσιάσετε τις συνέπειες του πιο θετικού μοντέλου, ποιο είναι το πιο ευνοϊκό σενάριο σε σχέση με τις συνέπειες, ε, ώστε ε, να επωφεληθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση από μια συμφωνία Brexit. Ποια κατά τη γνώμη σας, ποια κατά τη γνώμη σας είναι το ευνοϊκότερο σενάριο. Yes, I will, uh, very... Ναι, πολύ ευχαριστώ. Το απλούστερο, να το πω αλλιώς, ο τρόπος που έχουμε για να διατηρήσουμε μια κατάσταση συγκρίσιμη με αυτό που έχουμε τώρα είναι η διατήρηση της συμμετοχής στον ΕΟΧ. Δεν μιλώ για πολιτικές εκδοχές, μιλώ μόνο για την τεχνική ευκολία. Και γιατί, γιατί ήδη ε, καθώς έχει προϋπάρξει η ε, συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορεί να παραταθεί, να μετατραπεί σε μια συμμετοχή των νεόχων ή να περιοριστεί σε μια συμμετοχή στον Στο θέμα αυτό είναι νομοτεχνικά ακόμα ασαφές το αν θα πρέπει να γίνει μια ρητή εισδοχή στον νεόχων ή αν παραμένει μετά την αποχώρηση του Ρωμανόμενου Βασιλείου. Εν πάση περιπτώσει όμως για μας και για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν έχει μεγάλη σημασία γιατί παραμένει κανείς de facto σαν ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν είναι στο ΕΟΧ. Ε, αποχωρώντας λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον για τα θέματα αυτά θα διατηρούσε την ε, ε κατάσταση όπως έχει αυτή τη στιγμή. Η δεύτερη καλύτερη πρόταση θα ήταν ε, αν όχι ΕΟΧ, ΕΖΕΣ, ε, επιλογή η οποία θα έδινε μια προτεραιότητα στη συνεργασία, ειδικά για το τομέα των οπτικοακουστικών, εφόσον αυτό θεωρηθεί ιδιαίτερη σημασία. Φερρυπίν θα μπορούσαμε να εξεταστεί τι είδου συγκεκριμένη ειδική συμφωνία θα μπορούσε να ταθεί σε ισχύ προκειμένου να διαφυλαχθούν συνθήκε συνεργασία αντιστοιχέ με αυτέ που έχουμε τώρα. Δεν θεωρώ πάλι δύσκολη μια τέτοια επιλογή. Ε, Δεδομένου ότι διαφυλάσσεται το επίπεδο του κεκτημένου που έχει μέχρι τώρα επιτευχθεί και δεν βλέπω γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο. Ε, ωστόσο η εμπειρία που έχουμε από το ελβετικό μοντέλο δεν ήταν ε, απρόσκοπτη. Άρα Μα ενδιαφέρει να μπούμε σε ένα τέτοιο μοντέλο και αυτό δεν αφορά μόνο τα οπτικοακουστικά του δικό μου τομέα αλλά ε, γενικότερα γιατί εδώ έχουμε μέσα στον ΕΖΕΣ δύο επίπεδα συμμετοχή, δύο διαφορετικέ κατηγορίε μελών και ίσως αυτό δεν είναι το επιδιωκόμενο. Άλλη επιλογή, μια ε, συνεργασία τύπου εμπορικών συμφωνιών. Και εδώ διστάζω περισσότερο γιατί βεβαίως μπορεί κανείς να ε, συνάψει μια συμφωνία για μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών σε οποίο τομέα επιθυμεί. Αλλά αν δούμε τον, τομέα, ε, τον αντίστοιχο τομέα που αναπτύχθηκε στη συμφωνία με την Ιαπωνία, καταρχάς δεν κλείνει μια τέτοια συμφωνία μέσα σε ένα εξάμεινο και δεύτερον, εάν πρέπει να δούμε όλους τους τομείς που θα ανοίξουν σε μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, προφανώς δεν θα έχουν προτεραιότητα τα οπτικοακουστικά. Εμείς θέλουμε βέβαια τη συνεργασία με τον Ηνωμένο Βασίλειο και τα λοιπά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην όμως σε μια γενική προσέγγιση για μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, αυτό στο τομέα των οπτικοακουστικών δεν θα έχει την προτεραιότητα. Για να το πω διαφορετικά, ε, δύσκολα μου φαίνεται να αποκλίνει κανείς από τον μέχρι τώρα αποκλεισμό από συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών ε, του τομέα των, ε, του πολιτισμού ακριβώς επειδή έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Με τα φερσιμότητα μπορεί Φερρυπίν να περάσει, δηλαδή να αν, παραχθεί ο κανονισμός της μεταφερσιμότητα των ε, συνδρομών που έχουμε παραδείγματι και για τις διακοπές μας κλπ. Είναι κάτι το οποίο μπορεί σε μια πλήρως ε, ολοκληρωμένη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών ε, να περάσει. Ε, άλλοι τομείς όμως δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο εύκολο. Αλλά και πάλι θα έχουμε θέματα με, τη, με τα δικαιώματα πνευματικής διοκτησίας. Κυρία Τρίπλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κόλ. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Πριν από λίγα χρόνια όταν συζητούσαμε πάλι για την AVMS είχαμε συναντηθεί και είχαμε συνομιλήσει. Σας ευχαριστώ πολύ που μας εξηγήσατε τα διάφορα σενάρια ξεκινώντας από το καλύτερο σενάριο, δηλαδή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, που θα σημαίνει ότι <clears throat> ακόμα και αν γίνει το Brexit με μια ασυνθήκη άλλα Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει πολύ κοντά μας. Δεν θα είναι τέτοια μεγάλη καταστροφή. Εγώ βέβαια θα προτιμούσα χίλιες φορές να επανέλθουν ε, ε, σε δημοψήφισμα και να διαλέξουν την καλύτερη λύση οι άνθρωποι. Πάντως, θα το δούμε πάλι. Μου φαίνεται ότι όμως το εργατικό κόμμα δεν θα βοηθήσει σε μια τέτοια λύση. Αν κατάλαβα καλά τώρα, είπατε ότι σε κάποιο βαθμό πέραν Τη πολιτική συζητήσεως και του αφηγήματο υπάρχουν και οικονομικά συμφέροντα. Υπάρχει οικονομικό συμφέρον δηλαδή των ε, βιομηχανιών των media companies ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και των επιγραμμικών πλατφορμών έχουν το συμφέρον δηλαδή να παραμείνουν μέσα σε αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο που τους προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Είπατε ότι για το copyright τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, αλλά για κάποια για κάποιους από τους άλλους κανονισμού έχουν συμφέρον να μην αποχωρήσουν οι πλατφόρμες κλπ. Αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν δύο επίπεδα. Έχουν δηλαδή το πολιτικό επίπεδο που όλοι λένε «Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μεγάλη ανοησία. Από την άλλη μεριά όμω ε, υπάρχουν κίνητρα για να παραμείνουν. Διότι είναι ζητήμα, ζητήματα αγορά και ανάπτυξη αγορά. Ακόμα και για τι επιγραμμικές πλατφόρμες γιατί είπατε η αξιοπιστία και τα λοιπά των πλατφορμών είναι η τάση αυτή να έχουν δηλαδή καλή ρύθμιση στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί αν αληθεύει ακόμα και αν έχουμε α, πολλές αναταράξεις στο πολιτικό επίπεδο ίσως η επιρροή της αγοράς σε αυτή τη ε, ε, ε, δημιουργική βιομηχανία θα παραμείνουν, θα θελήσουν να παραμείνουν σε ένα πλαίσιο ε, πολιτικής ε, ρύθμισης διότι είναι προς το συμφέρον τους και τους προσφέρει πλεονεκτήματα. Ε, ρωτώ εάν είναι πράγματι έτσι, ότι δηλαδή έχουν ένα ενδογενές ας πούμε συμφέρον να μην αποχωρήσουν. Ναι, καλά το καταλάβατε. Βεβαίω εν μέρη είναι και κερδοσκοπικό. Πάντως για τον τομέα το broadcasting, έτσι νομίζω ότι είναι. Ας πάρουμε την, ε, το, την μεθοδολογία συμψηφισμού αδειών. Έχει, μπει, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για την εφαρμογή της ε, οδηγίας για την δηλώση ε, χωρίς σύνορα μαζί με την ΚΑΠΣΑΤ. Γιατί εάν εποφελούνται από την ιδέα τη χωρί αδειών. Δηλαδή ότι όταν είσαι εγκατεστημένο σε μια χώρα μπορεί να μεταδίδει σε όλε τι άλλε. Αυτό όμω δεν είναι όλη η υπόθεση γιατί είναι copyright clearance, δεν μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό έχετε μετά η οδηγία CAPSAT για ένα είδο τεχνολογία. Εκεί διευκρινίστηκε το θέμα αυτό. Και για να μπορεί ένα broadcaster να έχει τη νομική βεβαιότητα ότι εάν έχω ξεκαθαρίσει τα δικαιώματά μου στην χώρα που έχω την έδρα μου με προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε είμαι εντάξει αυτό νομίζω είναι ένα συνολικό πακέτο το οποίο τους ε, προσελκύει, δηλαδή τους παρακινεί να είναι μέσα και περισσότερο και όχι έξω. Τώρα, κάποια πράγματα ίσω είναι πιο ενδιαφέρον να μην τα έχουν, για παράδειγμα ορισμένες ποσοστώσεις. Η πραγματικότητα όμως είναι πάλι για τον τομέα broadcasting ότι πληρούνται οι ποσοστώσεις. Υπάρχει δηλαδή αρκετό περιεχόμενο που παράγεται ώστε να είναι προ το συμφέρον του να τα περιλαμβάνουν. Τώρα, οι ορισμένα επιμέρου κανάλια ίσω αυτό να μην συμβαίνει. Αλλά συνολικά πάντω η αγορά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τι παραδοσιακέ υπηρεσίε broadcasting και video on demand, υπάρχουν λόγοι να παραμείνουν. Τώρα, για τι πλατφόρμες video sharing, τα πράγματα εκεί είναι λίγο περισσότερο ε, περίπλοκα. Διότι εκεί έχουμε αρχίσει και επιβάλλουμε υποχρεώσει, πολύ σύντομα τουλάχιστον θα αρχίσουν να εφαρμόζονται οι υποχρεώσει μέσα στα πλαίσια τη AVMST και ίσω να μην είναι τόσο ελκυστικό για αυτές τις πλατφόρμες. Γιατί λέω όμως ότι μάλλον θα μείνουν. Διότι υπάρχει η ιδέα αυτή της δικαιοδοσία ότι αν δηλαδή έχεις, είσαι συνδεδεμένος με μια χώρα μέλος και, λέει, και λέω θα ήθελα ούτως ή άλλως να είμαι μέσα στη δικαιοδοσία μιας χώρας μέλους, τότε ίσως να προτιμήσουν να είναι ασφαλής, να είναι ασφαλής ότι είναι μέσα στη δικαιοδοσία αυτή, ότι συμμορφούνται δηλαδή με τις ρυθμίσεις. Και πάλι, εάν αποφασίσει η πλατφόρμα ότι θέλει να ακολουθήσει διαφορετικά μοντέλα, είναι τόσο ελκυστικό να αναπτύξουν ε, λύσεις software ώστε να έχουν μια διεύθυνση στην Ευρώπη με γεωγραφικό αποκλεισμό κλπ. Θα πούνε ότι η Ευρώπη, θα τη θεωρήσουν την Ευρώπη σαν έναν ε, νομικό χώρο όπου ε, θα αναπτύσσουν τα προϊόντα τους με τον ίδιο τρόπο. Αν δεν συμβεί αυτό, εάν υπάρξει μια μαζική κίνηση όπου όλες οι πλατφόρμες φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς καμία διασύνδεση με χώρες μέλη, δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ ενταγμένες σε πολλές από τις χώρες μέλη οι επιχειρήσεις αυτές. Δεν νομίζω δηλαδή να φτιάξουν βαλίτσες και να σκορθούν να φύγουν. Ευχαριστώ πολύ. κύριε Μπίλτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έφτασε κάπως ε, καθυστερημένα, λυπάμαι γι' αυτό, αλλά διάβασα τη μελέτη. Το 2017 ε, η σκαταλωθιακή θηρίδα Independent μιλούσε για τις καταστροφικές συνέπειες του Brexit ε, στη Βρετανική οπτικοακουστική βιομηχανία. Βέβαια, με αυτό που ακούσαμε δεν βλέπαμε πολύ αρνητικά θέματα. Για παράδειγμα, οι Βρετανικές ταινίες θα υπόψη στι ποσοστώσεις των ευρωπαϊκών έργων μια και εσεί επικεντρώνεστε στα νομικά ζητήματα, το θέμα της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου σε κάποια προγράμματα, όπως ε, το πρόγραμμα τη Δημιουργική Ευρώπη, ε, δεν ε, αναφέρθηκε. Εγώ ως Γαλλίδα δεν έχω συμφέρον να ταχθώ υπέρ της χρηματοδότησης των Βρετανικών προγραμμάτων και σχεδίων. Βέβαια, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι συνέβαλαν σε ταινίε όπως η ομιλία του Βασιλιά που είχαν παγκόσμια επιτυχία. Ε, τώρα θα ήταν παράλογο ε, οι Βρετανοί να ε, εκπίπτουν ε, τις συνεργασίες ενώ χώρες όπως το 25 συμπεριλαμβάνονται. Ευχαριστώ. Ποια είναι η γνώμη σας? Λοιπόν, βλέπουμε ότι το ζήτημα του Δημιουργική Ευρώπη, το πρόγραμμα και άλλα δεν τα έχουμε καλύψει από την έκθεση, γιατί εμείς είχαμε εντολή να εξετάσουμε το νομικό πλαίσιο μόνο. Αλλά όπως είπα και από την αρχή, έχει σημασία το γεγονός και δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι έχει μεγάλη σημασία ως ε, χώρος παραγωγής, ως τόπος παραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο και πρέπει να κοιτάξουμε αν έχει, αν έχει συμφέρον η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαρρήξει τους δεσμούς. Εξ αρχής είπα όχι. Το περιεχόμενο το οποίο παράγεται εκεί και η διάδοσή του στην Ευρώπη έχει πολύ μεγάλη αξία. Η ελεύθερη λοιπόν ροή πληροφοριών προηγείται της ιδέας της δημιουργίας μιας οδηγίας μέσα σε μια ενιαία αγορά. Η ιδέα δηλαδή της ανταλλαγής και του μοιράσματο πληροφοριών και ιδεών. Όσο πιο πολύ εισρωή στοιχείων έχουμε από το Ρωμανό το Βασίλειο, τόσο το καλύτερο. Επομένω, το συμφέρον δεν είναι μονόπλευρο. Τώρα, εάν αυτό μπορεί να καλυφθεί μέσα από συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδότηση στο μέλλον, εάν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει την συνεχιζόμενη ε, συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδότησης, τότε θα πρέπει αντίστοιχα όμως αυτό να συνοδεύεται και από την υπαγωγή στο διατακτικό τμήμα των νομοθετημάτων. Ή μπορεί κανείς να πει ότι προς το συμφέρον αμφωτέρων των πλευρών είναι να διατηρήσουν μια στενή συνεργασία. Και πάντως ε, η παραγωγή περιεχομένου και ο σχετικός κλάδος ε, δεν πρόκειται να μετατοπιστεί ε, με τη μια ε, από το Ηνωμένο Βασίλειο στην υπηρετική Ευρώπη. Θα ήταν λάθος να περιμένει κανείς κάτι τέτοιο. Ε, από την άλλη αυτό δεν θα με ανησυχούσε τόσο γιατί εδώ επανέρχεται η σημασία του, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ε, τηλεόραση πέραν των συνόρων, γιατί επιτρέπει τη διατήρηση ενός καθεστώτος, ακόμα και αν δεν υπάρξει συμφωνία, γιατί μπορούν στα ευρωπαϊκά έργα να συμπεριλαμβάνονται και οι βρετανικές παραγωγές, είτε έχουν χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια, είτε όχι. Ευχαριστώ. Και έχω και εγώ μια-δύο ερωτήσεις. Και η Ελίκα μετά θα πάρει το λόγο γιατί πολύ σωστά είπατε ότι σε κάθε διεθνή εμπορική σύμβαση και εμεί ω Επιτροπή Πολιτισμού ιδιαίτερη σημασία πάντοτε αποδίδουμε στο θέμα αυτό, τη συμπερίληψη δηλαδή των οπτικοακουστικών. Ε, τώρα ας πούμε ότι θα υλοποιηθεί το χειρότερο σενάριο, ότι δηλαδή περνάμε σε μια κλασική σύμβαση, συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο και τότε γιατί αυτό θα αποτελούσε ε, ρήξη σε σχέση με την μέχρι τώρα στάση μας ε, του αποκλεισμού δηλαδή των οπτικοακουστικών από τις συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών. Εάν ξεκινούσαμε λοιπόν με αυτή την αλλαγή στάσεις και επιλογών, τότε μήπως ανοίγαμε και τον ασκό του εόλου για κάθε μεταγενέστερη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. γιατί η Φερρυπίνη μπορεί να ανοίξει θέμα συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τι ΗΠΑ για άλλη μια φορά. Προ το παρόν δεν είναι ορατό κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορούμε και να το αποκλείσουμε. Οπότε θα ήταν πολύ δύσκολο να επιχειρηματολογούμε λέγοντα ε, σε μελλοντικέ συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών ότι να, για το Ηνωμένο Βασίλειο κάνουμε αυτή την ε, εξαίρεση τη εξαίρεση του αποκλεισμού, αλλά για τι άλλε έχουμε σοβαρά επιχειρήματα. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να προβάλλουμε σοβαρά επιχειρήματα και να ε, αλλάξουμε αυτή την πορεία. με την επιχειρηματολογία που έχουμε μέχρι τώρα. Και επίσης, Βέβαια, το καλύτερο θα ήταν να μην έχει αλλάξει τίποτα, αλλά το δεύτερο, θα ήταν, το δεύτερο καλύτερο θα ήταν η συμμετοχή στον ΕΖΕΣ πολύ καλά, δεν θα είχαμε στον ΕΟΧ, γιατί εκεί πέρα δεν θα είχαμε προβλήματα σε σχέση με την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τότε θεωρείτε ότι και με όλες τις άλλες μορφές συμφωνιών που απαριθμίσατε θα προχωρούσε στην υλοποίηση των οδηγιών ε, για τα οπτικοακουστικά του Ηνωμένου Βασίλειο. Δηλαδή θα έπρεπε να τις ενσωματώσει ως εθνική νομοθεσία ή θα έλεγε Φερρυπίν ότι παρότι δεν τον σωματώνουμε ε, γιατί το απαιτεί αγορά, περίπτωση κατά την οποία όμως θα μπορούσε να κάνει επιλεκτική εισαγωγή της, ε, των σημείων που την συμφέρουν για να έχει φερειπίν την πρόσβαση στην αγορά αλλά όλα τα άλλα σημεία τα οποία δεν θεωρεί τόσο, τόσο βολικά το ΕΒ Βασίλειο να τα άφηνε εκτός ε, της εφαρμογής στο εσωτερικό δίκαιο. Ή να πει όχι δεν με ενδιαφέρει καθόλου κάτι τέτοιο. Τι συνέπειες έχει κάτι τέτοιο για την αγορά. Όπως θέλετε. Καλώς. Λοιπόν, πολύ σύντομα στα γερμανικά για να απαντήσω. Ε, η πρώτη ερώτηση παίρνει την απάντηση που έδωσα και νωρίτερα ότι θα σήμαινε σημαντική απόκληση από τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Από την άλλη, βέβαια, θα μπορούσε να είναι μια μεμονωμένη περίπτωση σε μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών κανονικά ε, μιλούμε για διακεκριμένες αγορές και συζητούμε πού μπορούμε να τις ενώσουμε. Οπότε, προφανώς, εκεί δεν ξεκινούμε από τον τομέα των οπτικοακουστικών. Ίσως από την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων ή κάποιων συγκεκριμένων αγαθών. Όταν όμως έχουμε την αντίστροφη περίπτωση, δηλαδή ξεκινούμε από μια πλήρη ε, συμμετοχή σε μια εσωτερική αγορά, τότε και αυτό είναι και ζήτημα ε, που μπορεί κανείς να επικαλεστεί ως προηγούμενο ότι έχει νόημα να διαφυλαχθεί ένα κεφάλαιο ε, στα οπτικοακουστικά, το οποίο κανονικά δεν θα έμπαινε σε μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, χωρίς αυτό όμως να μπορεί να θεωρηθεί ως προηγούμενο και μια συμφωνία αντίστοιχη με την ε, Νότια Αφρική, επί παραδείγματι ούτε θα μπορούσε να αποκλειστεί το λοτομία των οπτικοακουστικών. Και μετά υπάρχει και το ερώτημα γιατί έχουν αποκλειστεί τα οπτικοακουστικά για πολύ ευλογέ αιτίε, γιατί δεν μπορούν να θεωρηθούν ω τα κοινά αγαθά ή εμπορικά προϊόντα και γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν σε κάθε ε, συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Θα έχει δηλαδή νόημα να διαφυλάσσονται, να παραμένουν χωριστά από άλλες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, γιατί έχουν τα ιδιαίτερά τους χαρακτηριστικά τα οποία διατηρούνται. Αλλά όπως είπα, στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου υπάρχουν σαφή επιχειρήματα πως είναι μια μοναδική περίπτωση. Δεύτερο, Ο κλάδος πιστεύω έχει ιδιαίτερο συμφέρον για αυτό το Communications Act και την διαφύλαξη του, την διατήρηση δηλαδή της ε, ισχύω του μέχρι τώρα, έτσι ώστε να μην ανατραπεί οτιδήποτε ή να μην εγκαταλειφθεί οτιδήποτε έχει μέχρι τώρα εξασφαλιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγματι, Δεν νομίζω ότι θα ήταν ελκυστικό για κανένα να απαλληφθεί αδίποτε διάταξη σχετική με τη διαφήμιση, Φερρυπίν. Ε, το θέμα είναι στις νέες διατάξεις τι γίνεται, τι θα ισχύσει. Εδώ η απάντηση είναι ότι εάν εξασφαλίζουν την πρόσβαση με ίσους όρους στην εσωτερική αγορά, τότε πρέπει η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο να γίνεται λέξη προς λέξη. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, τότε προφανώς υπάρχουν επιχειρήματα για το Ηνωμένο Βασίλειο να πει ότι δεν έχω την ε, χώρα εφαρμογή στην αρχή της ε, χώρας προελεύσεως. Και άρα έχουμε μια διαφορετική εφαρμογή. Εάν πει όμως ότι πρόκειται για μια διμερή σύμβαση, τότε μπορεί να έχει μια διαφορετική ρύθμιση. Ιδάλλως θα πρέπει να ισχύει ο κανόνας της χώρας προελεύσεως. Εάν όχι, ο κίνδυνος είναι να υπάρχει αυτή η επιλεκτική εφαρμογή που αναφέρατε, ε, όπως για παραδείγματι ε, με αποκλεισμό του παρόχου, των ESB. Και μετά ανοίγει όλο το θέμα του αν οι πλατφόρμες ε, καλύπτονται από τη ρύθμιση κτλ. Από την άλλη, εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να προχωρήσει λέγοντας ότι α, στη διάταξη για την τοποθέτηση, διαφημιστική τοποθέτηση προϊόντων κρατάω μόνο το 50% της διάταξης και το υπόλοιπο όχι. Όχι, κάποιοι τομείς από τις ρυθμίσεις θα βγουν ε, εάν πρόκειται να βγουν από την ε, διάταξη. Αναλόγως του προορισμού της προσφοράς και πάλι θα υπάρχει μια προσαρμογή στην ε, εγχώρια αγορά, αλλά υπό κάποιες γενικές ε, αρχές, κάποιους γενικούς κανόνες. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να αποκλείσει κάποια διαφοροποίηση ως προς την, διακοπέ ε, τις διακοπές για διαφημίσεις Φερρυπίν, η οποία όμως θα σχετίζεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εγχώριας αγοράς. Αλλά, όπως είπα, με την προϋπόθεση ότι αυτό σημαίνει πως διατηρείται η πρόσβαση στην αγορά. Μέχρι το, οι μέχρι τώρα διατάξει εξακολουθούν να ισχύουν θεωρητικά, η δάλωση για τις νέες θα υπάρχουν διαφοροποίησεις. Χέλγα η κυρία πάλι. Για το τελευταίο που είπατε, ότι στο Ενωμένο Βασίλειο διεξάγεται συζήτηση για τη ρύθμιση των πλατφορμών και κατά πόσο θα ξεπεράσει το EVMS. Μπορείτε να εξηγήσετε περισσότερο. Στη Γαλλία δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όχι, δεν είναι διαφορετικά. Στην Ιταλία όμω είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να καταλάβω ακριβώ τι συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεύτερο. Άλλη ερώτηση. Κυκλοφορούν φήμες ότι έχει ήδη υπάρχει ένα έγγραφο, ήδη διαπραγματευμένο δηλαδή, και ότι για λόγους ε, ας πούμε πολιτικής η Τερέζα Μέη παριστάνει σαν να μην έχει κλείσει ακόμα. Αν το ήξερα, δεν θα ήμουν καν εδώ. Ε, όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό, απαντά ο καθηγητής Κολ. Ε, γνωρίζω λιγότερα από ότι εσείς. Έχω άλλωστε και το βρετανικό μου διαβατήριο. Το λέω ανεκδοτολογικά. Δεν έχω όμως περισσότερες ας πούμε επαφές ή γνώσει από τι διαπραγματεύσει από αυτέ που έχετε εσεί. Για μένα είναι σαφέ ότι κάτι διαπραγματεύονται πίσω από κλειστέ πόρτες. Είναι όμως μια κατάσταση ανησυχητική, α το πω έτσι. Από την σκοπιά του παρατηρητού δηλαδή. Και βέβαια για αυτούς που εξαρτώνται από την αγορά είναι καταστροφή. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω με ποιου ακριβώ έχω μιλήσει. Έχω όμως μιλήσει με πολλούς από αυτούς που είναι στην αγορά και οι περισσότεροι έχουν Plan B ήδη στα συρτάρια τους. Plan B όμως σημαίνει ότι υπάρχουν δαπάνες, κόστη, ότι ε, θα υπάρχουν και ε, θα υπάρχει και κόστος για το προσωπικό. Θα είναι δραματική η κατάσταση αν αναγκαστούν κάποια στιγμή να ανοίξουν τα συρτάρια τους και να βγάλουν έξω το εναλλακτικό σχέδιο, το Plan B. Τώρα αυτή είναι βέβαια πολύ προσωπική παρατήρηση δική μου. Δεν μπορώ να πω ότι είναι επιστημονικά θεμελιωμένη. Τώρα να κάνω μια διόρθωση. Δεν υπάρχει πολιτική συζήτηση ακόμα για την ρύθμιση των πλατφορμών. Όμω υπάρχει πίεση από την κοινωνία. Για παράδειγμα, το Carnegie Trust έχει αναθέσει μελέτη για social media platforms σχετικά με το ποιε ευθύνε θα πρέπει να φέρουν και θα πρέπει να αναλαμβάνουν όχι μέσα στο περιορισμένο πλαίσιο που κάναμε εμεί για την οδηγία, σε πολύ, σε πολύ ευρύτερο πλαίσιο. Αν αυτό τώρα θα επηρεάσει την πολιτική διαδικασία, αυτό δεν μπορώ να το πω. Ωστόσο, πριν από λίγα χρόνια, να μην το λησμονούμε, είχε, γίνει, είχε κυκλοφορήσει μια αρκετά ευρεία ιδέα, για παράδειγμα, για την απαγόρευση πορογραφικού περιεχομένου ε, και online. Ε, να, να, πάει, να γίνει πολύ ευρύτερο από αυτό που κάνουμε στο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ίσως έχουν ε, ε βγάλει ρίζες κάποιες ιδέες που ξεπερνούν και την AVMS και ESP. Ευχαριστώ. Τζούλι Ward. Συγγνώμη. Ε, είχα σηκώσει το χέρι πολύ νωρίτερα και νόμιζα ότι με είχες δει. Ε, Μαρκ, ξέρεις ότι ε, δίνω μάχη για να ψηφίσει ο κόσμος, ε, γιατί νομίζω ότι ε, δεν έχουν αντιληφθεί όλοι που βρισκόμαστε και είναι πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση και μιλούμε για ένα τεράστιο και πολύ σημαντικό κλάδο, όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για πολλούς νέους καλλιτέχνες. Εγώ εκπροσωπώ το Μάντζεστερ και την Βόρειο Ανατολική Αγγλία και νομίζω ότι το Μάντσεστερ έχει μεγάλη θέση στα οπτικοακουστικά και αυτοί που εκπροσωπούν ε, τον Brexit είναι αυτοί που διέδωσαν ψέματα και δεν βρίσκονται εδώ και συνεχίζουν ε, να λένε ψέματα. Και είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε από κάποιον εμπειρογνώμονα, από κάποιο ειδικό, από κάποιον που έχει ε, κάνει έρευνα και έχει εκπονήσει μια μελέτη και μπορεί να μας παρουσιάσει ένα ευρύ φάσμα σεναρίων που κανένα όμως από αυτά δεν θα μας κρατήσει στο ίδιο επίπεδο με το οποίο βρισκόμαστε σήμερα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα πάντως να ποτίσω φόρο τιμής όσους βρίσκονται εδώ, δίνουν το παρόν και μεριμνούν και νοιάζονται για το τι θα γίνει στο μέλλον με το Brexit. Έχουμε πολλούς Βρετανούς που εργάζονται σκληρά και είναι ντροπή και σκάνδαλο που αυτοί που προκάλεσαν τον Brexit απουσιάζουν από τη σημερινή μας συνεδρίαση. Ε, θορύβησε το σχόλιο σου για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα μπορείς να το αναπτύξει λίγο παραπάνω, παρακαλώ. Γιατί η Τερέζα Μέη αποφάσισε να μην μας κρατήσει εντός του χάρτη θεμελιώδων δικαιωμάτων. Δεν νομίζω όμως ότι ο λαός του Ηνωμένου Βασιλείου αντιλαμβάνεται τις συνέπειες που θα έχει μια έξοδος μας και από το χάρτη θεμελιώδων δικαιωμάτων. Ε, Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε από σένα που είσαι εμπειρογνώμονα πώ η απώλεια των θεμελιωδών δικαιωμάτων μπορεί να επηρεάσει και το συγκεκριμένο κλάδο των οπτικοακουστικών μέσων. Και όχι μόνο να επηρεάσει όσου απασχολούνται στον κλάδο, αλλά και το κοινό, το κρατήριο, γιατί το κοινό είναι οι πάντε. Οπότε πώ θα επηρεάσει κάτι τέτοιο τον απλό άνθρωπο, γιατί σίγουρα θα επηρεαστούν οι καλλιτέχνε, οι οργανώσει, οι πλατφόρμε, ο κλάδο των οπτικοακουστικών μέσων, γιατί ε, η συνεργασία είναι πραγματικά ο ευρωπαϊκός τρόπος. Ε, έτσι δουλεύουμε στην Ευρώπη με συνεργασία. Και αν θέλει κανείς να έχει ασκήσει επιρροή, θα πρέπει να βρίσκεται εδώ, να κάθεται στην Τράπεζα του Διαπραγματεύσεων, να δίνει μάχη υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου και του κλάδου, όπως κάνουμε εγώ και η Τζιλ, ε, σε όλες τις συζητήσεις. Αλλά μία έξοδος από το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων θα έχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα για όλους και θα ήθελα αυτό το σημείο να μου αναπτύξετε. Ευχαριστώ. Δεν θα μιλήσω γενικώ για την συνέπεια που θα έχει μια έξοδος από το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά η ιδέα της δημιουργίας μιας αγοράς που θα υπάγεται στην οδηγία και στη συμβάση του Συμβουλίου σημαίνει περισσότερο περιεχόμενο, περισσότερη πολυμορφία, πλουραλισμό, πολυφωνία και η ιδέα ε, της εξόδου από τη, της, η ιδέα της σύμβασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ακριβώς ε, μία ελευθερία έκφρασης ε, και πληροφορίας και αυτό δεν περιορίζεται σε μία και μόνο χώρα. Γι' αυτό και πρόβλεψη της δυνατότητας διάδοση περιεχομένου διασυνοριακά δεν είναι θέμα μόνο αγορών ή αγοράς. Παρόλο που, αν το κοιτάξουμε ιδιαίτερα, όντω είναι ένα τεράστιο κλάδο και έχει μια πτυχή θεμελιωδών δικαιωμάτων γιατί αφορά τη δυνατότητα πρόσβαση στην πληροφορία. Αλλά θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση να κρατήσει το Ηνωμένο Βασίλειο εντό του πλαισίου τη με κάθε μορφή. Γιατί ένα κίνητρο θα είναι να έχουμε ένα επιπλέον κράτος ε, που ε, θα μπορεί να ε, διαδίδει ελεύθερα το περιεχόμενο του και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι αρκετό κίνητρο και σίγουρα αν έχουμε στενή σύνδεση με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι προς το συμφέρον μας. Αυτό θα πρέπει να συνειδητοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα για, για θα έχουμε άμεση εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της σύμβαση κάποια στιγμή στο μέλλον ή τι συνέπειε θα έχει αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και από το χάρτη. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι η ιδέα τη συνεργασία, τη στενή συνεργασία, δεν έχει μόνο οικονομική διάσταση, αλλά και διάσταση υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι και οι δύο πλευρέ θα υποφαληθούν από τη συνέχιση τη συνεργασία. Η σύμβαση για την διασυνοριακή τηλεόραση έχει ξεχαστεί κάπω γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο έχει περάσει το επόμενο στάδιο στην οδηγία για τι υπηρεσίε οπτικοακουστικών μέσων. Αλλά με ένα Brexit ίσω επιστρέψουμε στην οδηγία στη, τηλεόραση τη διασυνοριακή. Γιατί εκεί υπάρχει δυνατότητα ε, τη ε, ελεύθερη ε, διάδοση του περιεχομένου. Χωρί όμω το μηχανισμό επιβολή όπω προβλέπει η οδηγία. Οπότε ό,τι συμφωνίες και αν βρείτε, δεν θα πρέπει να επικεντρώνεστε μόνο στην οικονομική πτυχή, αλλά να λαμβάνετε υπόψη και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σας ευχαριστώ θερμά για την ε, τόσο συνεργαστική πιστεύω συζήτηση, που δεν κλείνει βέβαια με τη σημερινή μας ε, συνεδρίαση, αλλά μάλλον θα μας απασχολήσει για καιρό ακόμα. Και όπου βεβαίως θα πρέπει να αναζητήσουμε στο προσεχές διάστημα την καλύτερη δυνατή λύση. Και αυτό νομίζω ότι θα είναι λιγότερο δύσκολο να πιστούμε εμείς από ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ότι είναι προς το συμφέρον του να διατηρηθεί αυτή στην συνεργασία γιατί μερικές φορές είναι δύσκολο να πιστούν ε, οι ορισμένοι ότι μια λύση είναι πιο λογική. Αλλά πάντως ε, θα τα ξαναπούμε. Η μελέτη σας, η έρευνά σας είναι μια καλή βάση, είναι ένα καλό έγγραφο που μπορούμε να δούμε την έκθεση των θετικών και αρνητικών συνεπειών ε, της ε, αποχώρησης του νομανού Βασιλείου και με τα διάφορα εναλλακτικά σενάρια. Σε ευχαριστώ θερμά. Μας δώσατε λίγο φως στο σκοτάδι της άγνοιας και ίσως να είναι και το φως στο τέλος της σύραγγας ε, που δεν βλέπουμε ακόμη. Μια αχτίδα όμως διαφαίνεται. Και παραμένουμε σε επαφή και γι' αυτό αλλά και για άλλα θέματα. Ευχαριστώ. Αγαπητέ φίλε Αγαπητές φίλες και φίλοι, τώρα θα προχωρήσουμε στο θέμα υπαριθμών 8, αλληλεγγύη και συμπερίληψη. Μια αποκλεισμό δηλαδή. Αξίε που είναι σημαντικέ όχι μόνο για εκείνε και εκείνου που χρειάζονται μια χείρα βοηθεία, αλλά συνολικά για την κοινωνία μα και ε, πολύ σημαντικά πράγματα. Συμπερίληψη σημαίνει και συμμετοχή συμμετοχή και πέρασμα από το να είναι κανείς έξω στο να συμμετέχει πλήρως στο κοινωνικό γίγνεσθε και να είναι ένα πρόσωπο πραγματικά ενταγμένο. Αυτά αποτελούν προκλήσεις για ολόκληρη την Ευρώπη. Να ανοιχθούν δηλαδή δυνατότητες για τους πολλούς, για τους πολλούς πρόσφυγες από χώρες που αντιμετωπίζουν κρίσεις, ε, συγκρούσεις κτλ. Πρόκειται για Ηράκλειο άθλο που θα επιτύχει μόνο εάν μπορέσουν να συνεργαστούν οι χώρες μέλη και ιδίως ε, εάν η κοινωνία των πολιτών αναδείξει αρκετούς ενεργούς ανθρώπους οι οποίοι να συμβάλλουν ώστε να επιτύχει η ενσωμάτωση, η ένταξη αυτή. Έχουμε κοντά μας ε, τους εταίρους του Boosting Individual Competencies και αυτό το ε, project προωθήθηκε από τον Έρασμο. Θα μάθουμε και για μια διαδικασία η οποία έχει δημιουργηθεί με συνεργασία μαθητών και αποτελείται και, και αποτελεί μάλλον μάλλον πρόκειται για ένα, μια εσάρπα ας πούμε, που έχει φτιαχτεί από ε, την ένωση κομματιών που έχουν φτιάξει οι μαθητές. Δεν μπορώ δυστυχώς να αποκαλέσω όλους τους συμμετέχοντες με τα ονόματά τους. Απευθύνω ωστόσο τον χαιρετισμό στον κύριο Πιέρ Καρολάτσι, της οργάνωσης Κρέτα Ντιουβαλέ από τη Γαλλία, η κυρία Σουσάνα Κριστοφανέλο από το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Πάντουα, η κυρία Τερέζα Καρασκάλ της οργάνωσης Φεντερασιών Colectivos de Ενηλίκων πάλι, της Βαλοκιντάτ, ελπίζω να μην ε, ε, προφέρα πολύ άσχημα τα ισπανικά αυτά, την κυρία Science από το σχολείο Όιχεν στην Γερμανία, που ανέλαβε και τον συντονισμό του έργου και την οποία έχω την ευχαρίστηση να καλωσορίσω εγκάρδια εδώ δίπλα μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας σήμερα στην ε, συνάντηση. Κυρία Ζάιενς χωρίς περαιτέρω λόγια, θα σας παρακαλέσω στα επόμενα ας πούμε 10 λεπτά να μας εξηγήσετε λίγο το ε, project αυτό το οποίο έχετε ε, αναλάβει και φέρει εις πέρας. Έχετε το λόγο. Με ακούτε? Ναι, ναι, θαυμάσια, θαυμάσια σας ακούμε. Αγαπητή κυρία Κάμερα Εύερτ, αγαπητές και αγαπητοί βουλευτές, λέγομαι Ελέν Σάιενς και είμαι επικεφαλής ε, του Συμβουλίου του ε, Σχολείου όχεν στην Γερμανία και έχουμε αυτό το project που λέμε Boosting Individual Competences, η πρόθεση δηλαδή των προσωπικών ε, ικανοτήτων ή δεξιοτήτων. Έχουμε την Τερέζα Καρασκάλ, ε, της Ισπανικής ε, ας πούμε συνιστόσα, ο Πιέρ Καραλογκή που είναι ε, ο Γάλλος φίλος μας. Ίσως είναι ακόμη πιο σημαντικό αυτό που κάναμε, διότι είμαστε μια μικρή οργάνωση. Έχει λοιπόν ε, μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που έχουμε κάνει. Θα ήθελα λοιπόν ε, να εκφράσω τις ευχαριστίες μας που μας δώσατε την ευκαιρία να σας ε, κάνουμε μια μικρή αναφορά για το τι πετυχαίνει το Strategic Partnership Project του χρηματοδοτήτα από τον Έρασμο και που έχουμε ολοκληρώσει εμείς. Τέσσερα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων που αντιμετωπίζουν καθημερινά παρόμοιες προκλήσεις ενσωμάτωσης και ένταξης. Από την αρχή της κοινή μας προσπάθειας αποφασίσαμε να αναλύσουμε τις ανάγκες των προσώπων που βρίσκουν ε, να είναι δύσκολο να ενταχθούν στην κοινωνία. Όλες και όλοι είχαμε ήδη σχετικές εμπειρίες με ανθρώπους αναλφαβήτους ή με πολύ χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Ω ενήλικο είναι πολύ δυσκολότερο να έχει κανεί πρόσβαση στην εκπαίδευση από την αρχή από παιδί. Προσπαθήσαμε να βρούμε απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις. Πρώτα, ποια είναι τα πρόσωπα εκείνα που χρειάζονται βοήθεια ώστε να ενσωματωθούν με επιτυχία το προφίλ των προσώπων αυτών, Ποιε είναι οι βασικές τους ανάγκες, ποια εργαλεία μπορούμε να τους προσφέρουμε για να διευκολύνουμε την ενσωμάτωσή τους. Οι έρευνες που κάναμε μας οδήγησαν στα εξή συμπεράσματα. Εύκολα συμπεράσματα. Τα πρόσωπα που χρειάζονται βοήθεια για την κοινωνική τους ένταξη ή ενσωμάτωση είναι άνθρωποι από όλες τις υπήρους. Έχουμε ανθρώπους από παντού στα σχολεία μας. Και μάλιστα και, και ντόπιου οι οποίοι είναι αναλφάβητοι, έρχονται δηλαδή είτε άνθρωποι οι οποίοι εγκατέλειψαν το σχολείο πρόωρα ή που δεν πήγαν ποτέ στο σχολείο. Και μιλώ ε, για παράδειγμα για πρόσφυγες που συχνά δεν έχουν απολύτως καμία ε, παιδεία. Άνθρωποι με κάποια αναπηρία που δεν τους επέτρεψε να επισκέπτονται τακτικά το σχολείο άνθρωποι με περιορισμένη γνωστική ικανότητα που καμιά φορά τους αποθαρρύνει και τους οδηγεί να καταλήψουν το σχολείο ε, πρόωρα. Οι βασικές ανάγκες των προσώπων αυτών που εντοπίσαμε είναι ε, χρειάζονται ένα σπιτικό και μια οικογένεια, ε, να βρουν μια δουλειά, να μπορέσουν να επιβιώσουν με επαρκείς πόρους και να λαμβάνουν φροντίδα υγείας. το εργαλείο που ε, αναπτύξαμε έχει ας πούμε γενικό χαρακτήρα, μπορεί να εφαρμοστεί παντού. Στις ε, διεθνείς, διεθνείς μας συναντήσεις συζητήσαμε εντατικά τι μπορούμε να προσφέρουμε στα πρόσωπα αυτά, στις ομάδες αυτές προσώπων για την κοινωνική τους ένταξη. Ήταν σαφές ότι χρειαζόμαστε ένα εργαλείο που να είναι, εργαλείο πάντα εισαγωγικών, εύχριστο. Οι κοινέ μας προσπάθειες στόχευσαν ιδίω στην πανευρωπαϊκή δυνατότητα χρήσης του πόρου αυτού που ε, δημιουργούσαμε. Του δώσαμε και όνομα στην αίτηση που υποβάλαμε. Είχαμε συζητήσει ήδη τι θέλαμε να κάνουμε, να έχει δηλαδή κάποιο νόημα. Και το είπαμε ορισμός των οικείων εκπαιδευτικών βημάτων για την διευκόλυνση της ένταξης. Ε, και στα αγγλικά αυτό δίνει τα αρχικά ντρέσφη. Μετά από την αξιολόγηση των διαφόρων εργαλείων που επεξεργαστήκαμε, εγκρίναμε το σχέδιο που υπέβαλαν οι Γάλλοι εταίροι μας τους επόμενους μήνες χρησιμοποιήσαμε και ε, κάναμε, ε, θέσαμε σε δοκιμασία με το εργαλείο αυτό στα, ε, στις οργανώσεις μας. Και στη βάση των αποτελεσμάτων του κάθε εταίρου κάναμε και τροποποιήσεις ώστε να φτάσουμε στην τελική μορφή του εργαλείου αυτού που υποβάλαμε ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που ελπίζω να σας έχει διαβαστεί και σε εσά. Ποιο είναι το βασικό μήνυμα του εγγράφου μας που περιλαμβάνει αυτό το τρέσιο. Και πρώτο πρώτο είναι ο σεβασμός. Θεωρούμε ότι η επιτυχία της ένταξης και ε, συμπερίληψης του προσώπου ε, εξαρτάται σημαντικά από τον σεβασμό. Σεβασμός που σημαίνει ότι κάποιος τον ακούει. Δηλαδή ένα είδος ακρόασης του προσώπου πέραν από προκαταλήψεις. Χρησιμοποίησαμε λοιπόν τον τρέσφι στο πνεύμα αυτών των πεπιθήσεων. Τώρα, στην πράξη τον τρέσφι. Α, μετά το πρώτο μέρος που αφορούσε την διάγνωση και μια αξιολόγηση προσωπική και επαγγελματική όπου συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόσωπο, το Ντρέσφι μας προτείνει έναν αριθμό ε, εργαλείων για παράδειγμα για την αξιολόγηση του επίπεδου χρήση της γλώσσας, των δεξιοτήτων και έτσι να μας επιτρέψει να φτιάξουμε ένα ε, χαρτοφυλάκιο για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η δουλειά μας με μετανάστες και αναλφαβήτους μας δείχνει καθαρά ότι όπου δεν κατανοούνται η ομιλουμένη γλώσσα και η γραπτή γλώσσα υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιηθούν άλλα συμπληρωματικά εργαλεία. Και γι' αυτό παρακαλέσαμε έναν ε, ε, φίλο μας, ο οποίος φτιάχνει καρτούνς, ε, φτιάχνει κινούμενα σχέδια, να φτιάξει τέτοια κόμικς τα οποία ε, και ο οποίος λέγεται σκητσογράφος σε σωστά ελληνικά, να κάνει τα σχετικά σχέδια. Με τα σχέδια αυτά, τα οποία μπορείτε μάλιστα να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας και μάλιστα δωρεάν, είναι πολύ χρήσιμα για να μπορεί να διδάξει κανείς τα διάφορα θέματα. Έρχομαι στο συμπέρασμα και εδώ θα ήθελα να πω ότι το Ντρέσφι είναι ακριβώς αυτό που λέει και το όνομά του, δηλαδή ένα εργαλείο για να επιτρέψει μέσω των κατάλληλων εκπαιδευτικών βημάτων και να διευκολύνει μάλλον την ένταξη στην κοινωνία. Αναλάβαμε πολλές δραστηριότητες στη διάρκεια αυτή. Ένα μας ε, συνεπήρε πολύ, διότι ήταν αυτή τι δημιουργία αυτή της εσάρπας ε, της αλληλεγγύης. Ίσως το βλέπετε στις ε, φωτογραφίες και μπορούμε να σας το δείξουμε στο τέλος. Πριν μιλήσω για αυτή την εσάρπα της αλληλεγγύης, να σας μιλήσω για διδακτικό υλικό, για ε, πόρους και παιχνίδια που χρησιμοποίησαμε μέσα σε αυτά τα χρόνια όπου ε, δημιουργούσαμε το project. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα του project και μπορείτε βεβαίως και να τα κατεβάσετε και να τα χρησιμοποιήσετε δωρεάν. Οι Ισπανοί εταίροι μας ξεκίνησαν την ιδέα αυτού του wandering scarf, δηλαδή της περιπατητικής εσάρπας. Τη στείλαμε σε όλες ε, τις χώρες και θα δούμε εν τέλει το αποτέλεσμα. Στην πρώτη μας συνάντηση στο Όλχινγκ αποφασίσαμε ε, να πλέξουμε ε, ε, κομμάτια πούμε, της εσάρπας που να είναι μικρά, 20 επί 20 εκατοστά, ώστε να φτάσουμε στα δύο μέτρα αναχώρα. Και αρχίσαμε να ε, συλλέγουμε το αναγκαίο μαλλί. Δεν ε, ξοδέψαμε δηλαδή χρήματα από το project για να αγοράσουμε το μαλλί, βάσει το έδωσαν. Θα δείτε μετά στις ε, φωτογραφίες πόσο μαλλί μπορέσαμε να μαζέψουμε στη χώρα μας και μετά και στις άλλες χώρες. Ε, στη συνάντησή μας που, α, με συγχωρείτε μια στιγμή, οργανώσαμε, οργανώσαμε και εργαστήρια για να ε, πλέξουμε αυτά τα κομμάτια της ΣΑΡΠΑΣ και με την ευκαιρία αυτή να διεξαγάγουμε και μια εκστρατεία κατά του ρατσισμού και της και υπέρ μάλλον της ανεκτικότητας απέναντι στον άλλο. Είδαμε όταν συνεδρήκαμε πια στην Πάντουα ότι τα τετράγωνα αυτά που είχαμε φτιάξει από μαλλί ήταν όλα παρόμοια και αντιληφθήκαμε ότι τα διάφορα σχέδια που είχαμε πλέξει λοιπά ήταν τα σύμβολα της πολυφωνίας αυτής που θέλαμε να δείξουμε και οπτικά συνδέσαμε τα πρώτα κομμάτια 2 μέτρων και φτάσαμε να έχουμε ένα μεγάλο ε, μήκος 8 μέτρων. Μετά η γερμανική ομάδα αποφάσισε να συνεχίσει το πλέξιμο και να συνεχίσει ταυτόχρονα την εκστρατεία κατά του ρατσισμού και υπέρ της ανεκτικότητας απέναντι στους άλλους. Στα μέσα του 2017 είχαμε φτάσει στα 16 μέτρα. 16 μέτρα. Κόψαμε μάλιστα ε, κομμάτια και εκεί προσθέσαμε ανάμεσά τους δηλαδή ε, συνθήματα. Όχι ρατσισμό στην Ευρώπη. Ε, μαζί κοινή προσπάθεια για ένα καλύτερο κόσμο. Παιδεία για όλους. Ας διδαχθούμε μεν από τους δε και άλλα σχετικά μηνύματα. Τον Ιούλιο 2017 οργανώσαμε μάλιστα ένα flash mob, δηλαδή μια αυθόρμητη ας πούμε διαδήλωση στο Όλχινγκ στην πόλη από την οποία προέρχομαι και ολοκληρώσαμε επιτέλους και την Εσάρπα η οποία είναι 18,6 μέτρα μακρά με από 280 ξεχωριστά τμήματα τα οποία έχουν πλέξει τόσα πολλά ξεχωριστά χέρια. Αυτό λοιπόν, αυτή η Εσάρπα της αλληλεγγύης είναι σύμβολο της ε, πολυφωνίας, της ποικιλία πολιτισμών και πλούτου στην Ευρώπη και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Δεν θα ήθελα να χάσω την ευκαιρία αυτή να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εταίρους μας, δασκάλους μας, τους ανθρώπους που μαθαίνουν κοντά μας και σε όλα τα πρόσωπα που μας βοήθησαν ε, με το project αυτό, το οποίο τελειώνει φέτος τον Δεκέμβριο. Διδαχθήκαμε πολλά ημένα από τους ΔΕ. Ε, περάσαμε στιγμές ε, ζεστής συντροφιάς αλληλεγγύης και κάναμε, φτια... κάναμε καινούριου φίλους. Αγαπητή κυρία Κάμερ Εύρετ, αγαπητές και αγαπητοί ευρωβουλευτές, επιτρέψτε μου να επισημάνω στην Επιτροπή σας κάποια γεγονότα τα οποία επηρεάζουν την πολυφωνία των έργων αυτών που χρηματοδοτεί ο Έρασμος και τις ε, ανταλλαγές καλών πρακτικών, αλλά με αρνητικό τρόπο. το γεγονός ας πούμε ότι ένα θεσμικό όργανο είναι υπεύθυνο για ολόκληρο ε, το, ολόκληρη την επιδότηση δεν είναι καλό. Χρειαζόμαστε χρειαζόμαστε αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαφόρων φορέων και αυτοί όλοι πρέπει να είναι αξιόπιστοι. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι διάφοροι εταίροι έχουν ήδη λειτουργήσει και εργαστεί σε τέτοια προγράμματα. Εγώ, α πούμε, του γνώριζα όλου του εταίρου μου. Εσεί, νομίζω, όχι, δεν, γνωρίζαμε, δεν γνωρίζονταν οι Ισπανοί. Ε, δεν γνωρίζαμε του Ισπανού. Το γεγονός ότι ένα άλλο γεγονός που επηρεάζει την επιλογή εταίρων είναι και η γεωγραφική κατάσταση, διότι υπολογίζονται οι αποστάσεις με τρόπο που σπάνια αποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όμως αυτές οι κανονιστικές ρυθμίσεις οδηγούν τους, τα θεσμικά όργανα να προτιμούν εταίρους οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε μεγάλες πόλεις με καλές μεταφορές. Εάν όμως οι θεσμοί με του οποίου θέλω να συνεργαστώ βρίσκονται αλλού, σε μικρότερε πόλεις ή ε, μέρη, έχω τη δυσκολία να έρθω σε επαφή μαζί τους. Για να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα τώρα. Ασφαλώς και θέλουμε να συνεχίσουμε με την στήριξη του έρασμος και θέλουμε να ξεκινήσουμε και νέα project. Πιστεύουμε στην Ευρώπη και όλες και όλοι μας Εργαζόμαστε για πολλά χρόνια ε, σε τέτοια έργα και θέλουμε να συνεχίσουμε γιατί είναι σημαντικά. Ελπίζω ότι αυτή η εσάρπα αλληλεγγύης ε, θα ε, την αντιληφθείτε ως ένα σύμβολο, ως ένα μήνυμα και σας ευχαριστούμε και πάλι που μας επιτρέψατε να προσέλθουμε ενώπιόν σα για να σα αναπτύξουμε το έργο μα και νομίζω ότι μπορώ να πω εξ, όλων, ονόματος όλων, όλων μας ότι επιστρέφουμε σπίτι μα με το καλό συνέστημα ότι η Ευρώπη μα στηρίζει. Uh, ε, καταρχάς ευχαριστώ θερμά για την εντυπωσιακή πιστεύω παρουσίαση του έργου σας, του κοινού έργου, που αποδεικνύει και τη σημασία του, εργα... του Erasmus Plus και πόσο σημαντικά έργα μπορούν να προκύψουν ακόμα και σε συνεργασία μικρότερης κλίμακας εταίρων. Δεν χρειάζεται να είναι πάντα μεγάλες οι οργανώσεις που βρίσκονται πίσω από τα προγράμματα αυτά συνεργασίας οι μικρότεροι εταίροι που όμως είναι παντού στην Ευρώπη και όχι συγκεντρωμένοι σε κάποια σημεία μπορούν να κάνουν πολύ καλά και σημαντικά έργα. Και θα ήθελα να εξηγήσω σύντομα γιατί είναι εδώ τα έδρανά μας στην πρώτη σειρά άδεια δεν έχει να κάνει η εικόνα που βλέπετε με το γεγονός ότι δεν θεωρούν σημαντικά τα έργα σας ή την ε, δουλειά στην Επιτροπή μας οι βουλευτές. Απλώς έχουμε δύο μεγάλες ομάδες ε, που σήμερα διεξάγουν τις, ε, τα συνεδριά τους, τα μεγάλα ευρωπαϊκά συνεδριά τους. Στο Ελσίνκι είναι οι εξωδημοκράτες μια μεγαλύτερη ομάδα, αλλά και η Άλντε, φιλελεύθεροι. Ε, έχουν ε, σε κάποια άλλη πόλη της Ευρώπης αντίστοιχα ένα συνέδριο. Η, βουλευ... η βοηθή όμως των βουλευτών και οι ε, συνεργάτες των διαφόρων πολιτικών ομάδων βρίσκονται εδώ, σημειώνουν και ενημερώνουν βεβαίως στη συνέχεια τους βουλευτές τους για το σημαντικό αυτό έργο που μας παρουσιάσατε. Σας ευχαριστώ θερμά λοιπόν που είστε εδώ όλοι εδώ σήμερα για την παρουσίαση του έργου και παρακαλώ, εάν υπάρχουν παρατηρήσεις ή ερωτήσεις, ο κύριος Δρογεύσκη. Σας ευχαριστούμε θερμότατα για την παρουσίαση που μας κάνατε. Περιμένω λίγο για να φορέσετε τα ακουστικά σας. Για να ακούσετε τη διερμηνία. Ευχαριστώ λοιπόν θερμότατα για την παρουσίαση που μας κάνατε. Και τέτοιου είδους προγράμματα, τέτοια επιτεύγματα είναι ένα ακόμη επιχείρημα για να συνεχίσουμε τη μάχη μας ε, για τα κονδύλια του έρασμος ε, που εξυπηρετούν ε, το σύνολο της κοινωνίας και προσπαθούν να περιορίσουν τις ανισότητες και τους αποκλεισμούς και εσείς είστε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της, του νοήματος που έχει αυτός ο αγώνας για τα κονδύλια του έρασμος. Και έχω μια ερώτηση ως προς την κλίμακα τέτοιων διαβημάτων. Τι θα πρέπει να κάνουμε για να έχουμε τακτικά τέτοια σχέδια και προγράμματα, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οι στόχοι που έχουμε θέσει και που έχετε θέσει κι εσείς ε, να ε, μην περιορίζονται μόνο σε συγκεκριμένες περιφέρειες ή να έχουν περιορισμένη κλίμακα, αλλά να, έχουν, ε, να επεκτείνονται σε ευρύτερη κλίμακα και να έχουν και μόνιμο αποτέλεσμα. Γιατί ε, τέτοιες εμπειρίες της δικές σας μπορούν να αποτελέσουν ε, βέλτιστη πρακτική και να γίνουν υπόδειγμα, παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες οργανώσεις, για άλλους φορείς, για, άλλα κέντρα και για άλλες δημόσιους φορείς, γιατί πιστεύω ότι οι ειδικέ εμπειρίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και από άλλους φορείς. Σας ευχαριστώ και πάλι θερμότητα, γιατί πιστεύω ότι είστε πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση. Vielen Σας ευχαριστώ, κυρία Τρούπελ και μετά κυρία Γουορτ. Ναι, ευχαριστώ πολύ Πέτρα και θέλω και εγώ να έκφρασω τις ευχαριστίες μου για την παρουσίαση. Πάνω απ' όλο για τη δουλειά σας, γιατί αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα του τι μπορεί να προσφέρει η κοινωνία των πολιτών και πόσο μπορούμε χάρη στα προγράμματα αυτά να εξασφαλίσουμε τη συνεργασία, τις επαφές. Άνθρωποι που συχνά δεν έχουν την ευχέρεια να συμμετέχουν και να συνεργάζονται ε, μπορούν να το καταφέρουν χάρη στα προγράμματα αυτά. Έχετε κάνει εσείς τόση καταπληκτική δουλειά εσείς ως πολίτες. Είναι αυτό που λέμε στην ιδιόλεκτό μας empowerment, δηλαδή δυνατότητα ε, που προσφέρεται στους πολίτες να αναπτύξουν τις ε, δεξιότητες τους, να κάνουν κάτι καλό, κάτι περισσότερο και να αναπτύξουν από κοινού τις, ε, τα έργα τους. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα πολλά έργα που έχουμε δει να φέρουν τόσο καλά αποτελέσματα στον τομέα μας και που κρίνουν στη τελευταία ανάλυση και την ε, ε, αποδοχή, τη θετική αξιολόγηση των έργων, γιατί βεβαίως ε, χωρίς συγκρούσεις τίποτε δεν μπορεί να υπάρξει, αλλά πρέπει ο τελικός απολογισμός να είναι θετικός, όπως βλέπουμε και εδώ. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια και πάλι, ε, πολύ τιμή η δουλειά που κάνετε και εύχομαι και στο μέλλον να έχουμε την ευκαιρία να δούμε σημαντικά και θετικά τέτοια έργα. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε αυτή η υποστήριξη, γιατί μονόδρομος ε, δεν είναι τίποτε και εμείς βεβαίως πρέπει να στηρίζουμε τα προγράμματα και να εξασφαλίζουμε την χρηματοδότησή τους για να προχωρήσουν, αλλά ταυτόχρονα πρέπει και οι πολίτες να αποδέχονται τα προγράμματα αυτά και να δέχονται τη χρηματοδότησή τους και να την προάγουν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ward, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε για την παρουσίαση αυτού του εξαιρετικού έργου που νομίζω αποτελεί και την, ε, το απάβγασμα των ευρωπαϊκών αξιών ε, για ολόκληρη την Ευρώπη εκφράζεται η υποστήριξη μέσω του Erasmus Plus στον άνθρωπο, γιατί η Ευρώπη κατά βάση είναι ένα έργο που απευθύνεται στον άνθρωπο και αυτό που μπορείτε να κάνετε σήμερα, αυτό που δείχνετε σήμερα εσείς, είναι το πώς μπορείτε να πλησιάσετε τον άνθρωπο και να του δώσετε την αξία του ως ανθρώπινου όντως μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Μ' αρέσει πολύ αυτή η ιδέα με το σάλι, με την εσάρπα, της αλληλεγγύης. Είναι εξαιρετική ιδέα, η αλληλεγγύη είναι το κύριο μας έργο νομίζω και το καθήκον μας και πολλοί το έχουν λησμονήσει αυτό γιατί η κρίση που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη δεν είναι κρίση μεταναστευτική, είναι κρίση αλληλεγγύης. Πρόσφυγες υπάρχουν και στο Λίβανο την Ιορδανία, από την Παλαιστίνη. Είναι πολλοί οι πρόσφυγες, ελάχιστοι αυτοί που φτάνουν ε, και διασχίζουν τα σύνορα των ευρωπαϊκών κρατών. Πρόβλημα λοιπόν είναι η απουσία αλληλεγγύης και ε, πιστεύω ότι θα πρέπει αυτό το έργο να ε, καταστεί πιο γνωστό, να διαδοθεί περισσότερο. Το λέω γιατί συχνά επισκέπτομαι κέντρα υποδοχής προσφύγων. Συναντώ πρόσφυγες και συχνά μου λένε «Ε, ναι, καλά, οι νέοι μόνο, η νεολαία μόνο ασχολείται με τους πρόσφυγες ή όλοι αυτοί που τρέχουν στα φεστιβάλ ε, δεξιά και αριστερά να ακούσουν μουσική. Αλλά βλέπω εδώ ακριβώς το αντίθετο, την απόδειξη του αντιθέτου. Βλέπουμε μια οργανωμένη, μια ολοκληρωμένη κοινότητα η οποία έρχεται να εκδηλώσει και αυτό με την παροχή της, ε, με την εκδήλωση της συμπόνιας ε, που οφείλουμε όλοι σε τελευταία ανάλυση και εδώ δεν είναι κάτι το οποίο ωφελεί μόνο τον πρόσφυγα ή τον μετανάστη. Σαφώς μας λέτε ότι όλοι όσοι έλαβαν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα κέρδισαν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι ήρθατε να μας παρουσιάσετε το έργο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ και εγώ θερμά για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Εξαιρετική δουλειά σας. Έμπρακτη η αλληλεγγύη που προσφέρετε μέσα από το έργο σας, η στράτευση όλων αυτών των ανθρώπων για να προσφέρουν. Και αυτό δεν είναι μόνο... Ε, το ότι καταφέρατε ένα πολύ καλό έργο να αναπτύξετε, αλλά ότι μπορέσατε να το συνδυάσετε, να το συνδέσετε με άλλα αξιόλογα έργα. Αυτό είναι το ε, πρόγραμμα Εράσμους. Αυτό προσφέρει ότι φέρνει κοντά ανθρώπους, ότι τους δίνει κίνητρα, ότι τους υποκινεί να δραστηριοποιηθούν, να στράτευθούν, να εργαστούν μέσα στις κοινότητές τους. Αισθάνονται έτσι όλοι ενωμένοι. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το όφελος από τέτοια έργα, από τέτοια προγράμματα. Για άλλη μια φορά λοιπόν, θερμές ευχαριστίες και από μένα. Η κυρία Μπίλτ όμως, ε, βλέπω να είστε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, κυρία μου, κύριε, ευχαριστώ πολύ. Είναι εξαφές ότι έχετε ετοιμάσει το έγγραφο αυτό για να ωφεληθούν στο δυνατόν περισσότεροι. Μας δίνει μια σαφή εικόνα των δραστηριοτήτων οργάνωση όπως η δική σας. Έχω λοιπόν την περιέργεια να μάθω περισσότερα και έτσι επισκέφτω επισκέφθηκα την ιστοσελίδα σας ε, για να ενημερωθώ ότι δραστηριοποιήστε σε, χώρες, σε τέσσερις χώρες, ε, Γερμανία, Ισπανία και ε, Ιταλία και Αγγλία. βλέπω όμως, ε, συγγνώμη και άλλη μία, ωστόσο βλέπω ότι χρησιμοποιείτε την αγγλική γλώσσα που δεν είναι καν επίσημη γλώσσα μιας από τις τέσσερις χώρες οι οποίες δραστηριοποιείστε, πράγμα το οποίο με εξαφνιάζει. Πώς είναι δυνατόν αφού η γνώση μιας γλώσσας, της γλώσσας της χώρας στην οποία βρίσκεται κανείς, έχει μεγάλη σημασία για την ενσωμάτωση. Εγώ που κατοικώ στη Λορένη της, Γερμανίας, της Γαλλίας ε, όμορης με την Γερμανία, ε, βλέπω ότι αρχίζουμε σιγά σιγά να εισάγουμε τα γερμανικά στα δημοτικά συμβούλια για να έχουμε καλύτερη συνεργασία με τους Γερμανούς γείτονες και εκείνη το αντίστροφο. Ε, αλλά ερωτώ, ε, κονδύλια. Τι κονδύλια παίρνετε στο πλαίσιο του Erasmus Plus. Δεύτερον, βλέπω ότι χρησιμοποιείτε μόνο τον όρο μετανάστες, ενώ νωρίτερα χρησιμοποιήσετε και τον όρο πρόσφυγες. Ερωτώ λοιπόν, Έχετε τη βεβαιότητα ότι βοηθάτε ανθρώπους που είναι νόμιμοι μετανάστες ή μήπως και αυτούς που παραβαίνουν τον νόμο. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω το πρόβλημα με την ιστοσελίδα σας μπορούμε να το συζητήσουμε. Ίσως είναι διαθέσιμο ε, και σε άλλες γλώσσες ή στο σελίδα. Ο κύριος Κόλος, όχι θα σας απαντήσω, το κείμενο είναι στα αγγλικά για σας, για να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση για όλους. Ωστόσο τα έγγραφα είναι αναλόγως της χώρας προσβάσιμα στα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά, αναλόγως της χώρας. Το δικό μας το κομμάτι έχει τα έγγραφά του στα γαλλικά, στη Γαλλία καθένας στη δουλειά του, ε, στη γλώσσα του εργάζεται. Για την άλλη σας ερώτηση... Ναι, κοιτάξτε, είμαστε όλοι, και αυτό θα απαντήσει και στον κύριο Στρογεύσκη, οργανισμοί είμαστε με δραστηριότητε κατάρτισης, ε, υποστήριξης εκείνων που έχουν ανάγκη από μια ε, στήριξη για να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Κατάρτιση, επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε όλοι, η καθημερινή μας δουλειά. Έτσι, συνοδεύουμε αυτούς τους ανθρώπους και τους εκπαιδεύουμε. Και το έργο, για να απαντήσω στον κύριο Στρογεύσκη, είναι επιπλέον ε, ένα μέσον επικοινωνίας μεταξύ μας επικοινωνίας, συνεργασίας και σχεδιασμού που δεν θα μπορούσε ο καθένα μόνο του να κάνει με τους εθνικού πόρου. Γιατί στη Γαλλία δεν υπάρχει χρηματοδότηση της, ε, του σχεδιασμού της κατάρτισης ή τη συνεργασίας με άλλους Ευρωπαίους εταίρους που θα μπορούσαν ε, όλα αυτά δηλαδή, μας επιτρέπουν να εξασφαλίσουμε νέες ιδέες, προτάσεις, ε, δημιουργία. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τη Γαλλία, σε όλε τι χώρε Σε καμία χώρα δεν υπάρχει χρηματοδότηση για τέτοιου είδου συνεργασία που μα εξασφαλίζει η Ευρώπη και το Erasmus Plus και έτσι είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Και η τελευταία ερώτηση από εσά εκεί. Είμαστε οργανισμοί με ε, δημόσια παρουσία ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και εργαζόμαστε στο πλαίσιο του νόμου. Καταρτίζουμε εκείνους που έχουν δικαίωμα στην κατάρτιση πρόσβαση στην κατάρταση. Είτε είναι στη Γαλλία, την Ιταλία κτλ. Ελεγκτέ δεν είμαστε, αλλά εργαζόμαστε πάντα στα πλαίσια του νόμου της επαγγελματική κατάρτισης στη Γαλλία ή αντίστοιχα στη Γερμανία, την Ιταλία που ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση, για τις απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ για το έργο σας. Συνεχίστε, σας ενθαρρύνουμε. Συνεχίστε, αναπτύξτε και άλλα τέτοια συναρπαστικά έργα και ε, συνεχίστε να δίνετε αυτό το θετικό παράδειγμα και σε άλλους που θέλουν να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε και πάλι θερμά. Τώρα θα θέλαμε πράγματι να δούμε αυτή την υπέροχη εσάρπα και να την ε, ανοίξουμε εδώ, να την δουν όλοι. Όλες και όλοι έλθετε εδώ μπροστά να μας δείξετε αυτό, αυτή τη θαυμάσια ε, Σάρπα ή Σάλι που ε, το βαφτίσατε Σάλι της ε, αλληλεγγύης.